Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο σημείο 26 ημέρες της διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την Vivian Redding, η οποία είναι ιδιαίτερα καλόδεκτη στην Επιτροπή μας για τα θέματα δικαστικών και εσωτερικών θεμάτων. Θέλουμε να οργανώσουμε τη συζήτηση και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε υποφελώ το χρόνο μας. Προβλέπετε να έχουμε τη συνεδρίαση αυτή μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την παρουσίαση των απόψεων της κυρίας Ρέντινγκ για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρόταση την έχει παρουσιάσει η Κομισιόν, την προστασία επίσης των προσωπικών δεδομένων και τον οδικό χάρτη για τη δικαστική συνεργασία. Θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και αν χρειαστεί άλλος ένας γύρος ερωτήσεων. Πρόκειται λοιπόν για μια συζήτηση η οποία, χωρίς αμφιβολία, θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Δίνω λοιπόν το λόγο, αφού την καλωσορίσω για μια ακόμα φορά, στην κυρία Ρέντι. Σας εύχομαι. Ό,τι θες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για την υποστήριξη προς τα θύματα εγκλημάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για το έργο το οποίο έχει γίνει από τη βάση της ε, νομοθετικής πρότασης, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί. Χάρη <clears throat> στην ιδιαίτερη προσήλωση του εισηγητού και του, των σχεδόν εισηγητών, έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό ο πρόεδρος Επιτροπής σας μου ζήτησε να αναφερθώ στην οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά για το θέμα της ενδεχόμενης υπάρξης ενός Γενικού Εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάω με τα θέματα και την πρόοδο που έχει γίνει στον αγώνα κατά των απατών και των αστασταλιών. Στι 11 Ιουνίου η Κομισιόν ενέκρινε μια πρόταση οδηγία, η οποία έχει σε στόχο να δώσει τα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αγωνιστεί εναντίον των απατών που πλήττουν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια προτεραιότητα όλων μα. Ιδιαίτερα μέσα στην τωρινή συγκυρία και τι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε όλοι, και στη στιγμή που είναι υποδιαπραγμάτευση το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η έκταση των παρανόμων δραστηριοτήτων που οδηγούν σε απώλειες του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντυπωσιακή. Υπάρχουν εγκληματίες που δίδουν λανθασμένες πληροφορίες θεληματικά για να πάρουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το 2010 τα κράτη-μέλη ανέφεραν περιπτώσεις απατών με συνολικό ύψος 600 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι μονάχα τα ποσά τα οποία αναφέρθηκαν. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι το πραγματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ακόμα και ένα ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων να πηγαίνει στα, στις τσέπες εγκληματιών. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τη χάνουν ομοιόμορφης προστασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι κανόνες ποινικού δικαίου των κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν απάτες προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εμβαλωματικοί. οι ποινές, οι κυρώσεις για το ίδιο αδίκημα ποικίλουν από πολλά έτη μέχρι ένα απλό πρόστιμο, μέχρι ακόμα και τίποτα απολύτως, δηλαδή έλλειψη αξιοπίνου. Και αυτό εξαρτάται από το μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται κανείς και αυτός είναι και ένας λόγος και ένα κίνητρο για τους ε, εγκληματίες να εκμεταλλευτούν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια βιώσιμη κατάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό ταμείο για να επενδύουμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για υποδομή, για να υποστηρίξουμε τους γεωργούς μας και 27 διαφορετικές προσεγγίσεις αν υπάρξει κάποια απάτη σε βάθος, σε βάθος αυτού του ταμείου. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια απλή λογική. Αν έχουμε ένα ομοσπονδιακό προπολογισμό με χρήματα τα οποία προέρχονται από του προλογούμενου 27 κρατών μελών, τότε χρειαζόμαστε επίση και ομοσπονδιακή νομοθεσία για την προστασία αυτού του προπολογισμού. Εάν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάρουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, κανείς δεν θα το κάνει για λογαριασμό μας. Όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικό από τα εγκλήματα τα οποία την χάνουν δίωξη σε εθνικό επίπεδο. Επομένω, η προτινόμενη οδηγία κατά των απατών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το κενό. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δίωξη και τον κολασμό αδικημάτων έναντι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται με τον τρόπο αυτό και με τους νέους αυτούς κανόνες οι εγκληματίες δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές στα νομικά συστήματα των κρατών μελών και δεν θα έχουν ασφαλή καταφύγια όπου μπορούν να κρυφτούν. Θα ήθελα τώρα να σταθώ λίγο σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία της πρότασής μας. Η πρότασή μας προτείνει κοινού ορισμού για αδικήματα κατά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απάτε και συναφή θέματα, κατάχρηση διαδικασιών διαγωνισμών, διαφθορά, ξέπλυμα χρημάτων, το λεγόμενο, ε, τις λεγόμενες περιστρεφόμενες πόρτες για το ΦΠΑ κτλ. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια, μια εναρμόνιση για ποινές από μήνες φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια για τα πιο σημαντικά εγκλήματα κατά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζημίες από, μέχρι, από 100.000 σε απάτες ή 30.000 και πάνω σε πλήσιμο χρημάτων. Επίσης, θα προτείνει χρόνους, περίοδο παραγραφής η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια δικήματα, γιατί σήμερα Αυτές οι περίοδοι παραγραφής είναι πάρα πολύ σύντομες και ουσιαστικά εμποδίζουν τις αρχές, τις ε, διοκτικές αρχές να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί στην δίωξη αυτών των εγκλημάτων. Τέταρτον, η πρόταση θα κάνει πιο εύκολο να ανακτήσουμε ποσά που έχουν τύχει απάτης, συνδέοντας αυτήν την ε, οδηγία με την οδηγία περί κατασχέσεως, η οποία είναι τώρα υπό εξέταση. Και φυσικά θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε μια πολιτική μηδενική ανοχή για τι απάτε κατά του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μπορεί να σα φαίνονται απόλυτα λογικά. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω στην Επιτροπή σας ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Γιατί βλέπω να υπάρχει κάποια διστακτική αντιμετώπιση σε ορισμένα κράτη-μέλη σε σχέση με ένα μηχανισμό που θα προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι εύκολη συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτα απαραίτητη. Γι' αυτό βασίζομαι σε εσά για να με βοηθήσετε σε αυτό το εγχείρημα. Δεύτερο σημείο, όπως ε, ενθυμίστε από την ομιλία του πρώτου της Κομισιόν που παρουσίασε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε την πρόθεση της Κομισιόν να καταθέσει μια πρόταση για τη δημιουργία ενός γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιπτώσεις απάτης που αφορούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οδηγία που ανέφερα προηγουμένως θα αναφέρει τους αρμόδιους ορισμούς και τις αρμόδιες κυρώσεις, όλα αυτά τα θέματα θεωρούνται πολλέ φορέ από του εισαγγελεί ω θέματα χαμηλή προτεραιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο οι συνεργάτε μου επεξεργάζονται μια πρωτοβουλία για να θεσπιστεί ένα γραφείο Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, Γενικού Εισαγγελέα, από τη βάση του άρθρου 86 των συνθήκων. Το γραφείο αυτό το εισαγγελικό θα έχει τη, δυνατότητα να ξεκινάει δίωξη σε όλα τα κράτη-μέλη και με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα έλθουν ενώπιον των δικαστηρίων αυτοί οι οποίοι διερευνούν απάτες. Επομένως δεν είναι όπως θεωρήσανε όλοι ένας συλλήβδεν γενικός εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απλώς ένας εισαγγελέα, ο οποίος θα συντονίζει το έργο των κρατών μελών στις περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε προς την εκκίνηση αυτού του εγχειρήματο. ώστε δεν μπορώ να σας πω από τώρα σε λεπτομεριακό επίπεδο πώς θα λειτουργήσει αυτό το εισαγγελικό γραφείο. Όπως όμως αναφέρεται στις συνθήκες, η αρμοδιότητα του θα εστιάζεται σε απάτες με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά η προετοιμασία, για τη δημιουργία αυτού του εισαγγελικού γραφείου θα εμπλέξουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν καιρό και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι είχα μία συνάντηση με τους εθνικούς εισαγγελείς και με την Eurojust ένα άλλο φορέα και με την Όλαφ. από το πολύ ταξίδι, θα ξεχνάω, με την Όλαφ, που είναι ένας από τους φορείς που πράγματι ζήτησαν να γίνει πραγματικότητα αυτή η εισαγγελική αρχή και όπως ε, έχω πει και στο παρελθόν, αυτό θα είναι μια μετεξέλιξη κατά κάποιο τρόπο στα πλαίσια του Eurojust. <clears throat> η δημιουργία αυτού της εισαγγελική αρχής θα σας κρατήσω εξάλλου ενήμερους για όλα αυτά τα οποία θα λάβουν χώρα. Δικονομικά δικαιώματα τώρα. Έρχομαι στο επόμενο θέμα. Το 2009 έχουμε θεσπίσει μία φιλόδοξη ημερήσια διάταξη ώστε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων την χάνουν εγγυήσεων. Θέλουμε κοινού κανόνε για να εξασφαλίσουμε ότι ο κοινό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνη, ο οποίο βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων, θα λειτουργεί ορθά. Γιατί χρειαζόμαστε ελάχιστου κανόνε για δίκαια δίκη που ενισχύει τα δικαστικά μας συστήματα. Χάρη στη δική σας συνεργασία έχουμε και δύο μέτρα τα οποία έχουν ήδη γίνει δεκτά. Το δικαίωμα στη μετάφραση και την ε, διερμηνία σε ποινικέ διαδικασίες και το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Τον Ιούνιο πέρσι παρουσίασε ένα τρίτο μέτρο το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο για μένα αποτελεί και τον πυρήνα των δικονομικών δικαιωμάτων και του συναφού οδικού χάρτη, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για το θέμα αυτό. Γιατί οι πολίτες μας θα πρέπει να έχουν επαρκείς διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε περιπτώσεις όπου κατηγορούνται ή θεωρούνται ύποπτοι για εγκληματικές ενέργειες. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ψήφο προσανατολισμού σας στις 12 Ιουλίου και την έκθεση της κυρίας Αντωνέσκου. Όλα αυτά με έχουν καθησυχάσει γιατί ξέρω ότι ήταν φιλόδοξο το εγχείρημα. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών δείξατε ότι πρέπει να θεσπίσουμε υψηλής ποιότητος πρότυπα στον τομέα αυτό, να διατηρήσουμε και να, να διατηρήσετε και να ενισχύσετε αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν και θέλω ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε υπογραμμίσει την πάρα πολύ σημαντική αρχή της εμπιστευτικότητας. Θα πρέπει να διέπονται αυτές οι διαδικασίες από εμπιστευτικότητα όταν κάποιος ο οποίος είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος επικοινωνεί με το δικηγόρο του. Θα πρέπει να υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες εξαίρεσης από αυτό το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικηγόρο και ιδιαίτερα στις χώρες όπου εκδίδεται ένα ένταλμα, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες σε περίπτωση παραβίασης αυτού του δικαιωμάτος. Του δικαιώματος. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνέσκου για την άοκνη εργασία της για αυτό το θέμα. Πριν από δύο εβδομάδες έγινε ο πρώτος τριγωνικός διάλογος σε επικοδομητικό πλαίσιο και κλίμα η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στο να μπορέσει να επιτύχει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της θητείας της Κυπριακής Προεδρίας και εγώ υποστηρίζω πλήρω αυτή την προσπάθεια και θα συνεργαστούν οι υπηρεσίε μου μαζί με την Κυπριακή Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτύχουν το στόχο αυτό. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι διαπραγματεύσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα απαιτηθεί περαιτέρω ευελιξία για να καταλήξουμε στη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των υπόπτων από τη μία και στις ανάγκες από την άλλη για μια ουσιαστική έρευνα και ανάκριση από την άλλη. Πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε οποιαδήποτε λύση στην οποία καταλήξουμε θα πρέπει να σέβεται και να ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το τελικό κείμενο, όποιο και αν είναι, θα πρέπει να δίδει τις κατάλληλες εγγυήσει έτσι ώστε τα δικαιώματα σε μια σωστή και δίκαιη δίκη ε, είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι μένει να κάνουμε λοιπόν ακόμα περισσότερο στον τομέα αυτό. Όταν μιλάμε για τα θύματα και σας ευχαριστώ Γι' αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο συνεργάζομεθα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με την Επιτροπή Γυναικών. Αυτό δείχνει πόσο μια από κοινού προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, στην περίπτωση των παιδιών που κατηγορούνται ας πούμε αυτόματα εντάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων. Προεβλέπεται δηλαδή και στα προηγούμενα μέτρα. Όλοι όμως αυτοί θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή διεξάγει μια μελέτη η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των επιπτώσεών της και προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τις συνέπειες που έχει η έννοια της ε, εκ των προτέρων θεώρησης ότι είναι αθώος ο κατηγορούμενος μέχρι τη στιγμή που θα δικαστεί. Έχουμε λοιπόν κάνει πολλά. Συνεχίζουμε την επεξεργασία του θέματος και τελικά οι νέες μας προτάσεις θα κατατεθούν. Να μου επιτρέψετε, Πρόεδρε, να θέσω τώρα ένα θέμα το οποίο η δική σας Επιτροπή έχει, με το οποίο η Επιτροπή σας έχει απασχοληθεί και μάλιστα χθε το συζητήσατε κιόλας σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Αναφέρομαι στο θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, η έκθεση τέθηκε, η μεταρρύθμιση αυτού του τομέα τέθηκε και ξεκίνησε τον μήνα Ιανουάριο. Είμαι ευτυχής σαν επίτροπος γιατί έχω πέσει πάντα σε πάρα πολύ αποτελεσματικούς εισηγητές. Ο κύριος Δρούτσας και ο κύριος Άλμπρεχτς κάνουν μια εξαιρετική δουλειά χωρίς αποκλισμούς. Έχουν κάνει εξαιρετικές διαβημένες διαβουλεύσεις έχουν υιοθετήσει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και λέω φιλόδοξο γιατί στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2013 μέσα στο 2013 μέχρι το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας. Με, ξέρω ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος αυτός, αλλά οι ρυθμοί με τους οποίους εργάζεστε το καθιστούν εφικτό. Ήδη τα πρώτα έγγραφα τα οποία ε, πρότειναν ε, οι εισηγητές έχουν ενδιαφέρον. Προτείνω ότι οι δύο προτάσεις μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα. Συμφωνώ με την αντιμετώπιση του θέματος σαν πακέτο, το θεωρούμε αυτό βασική προϋπόθεση. Είδα τους τομείς στους οποίους πιστεύουν οι δύο εισηγητές ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις και συμφωνώ και θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσω ότι στο άτυπο συμβούλιο του μηνός Ιουλίου, που πήγατε και εσείς μέρος πρόεδρε, ε, ήδη τέθηκαν κάποια θέματα όπως οι εφαρμοστικές πράξεις, ε, η κατεξουσιοδότηση πράξης, τα γραφειοκρατικά θέματα, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι έχει συντελεστεί κάποια πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς. Έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η αρχή ότι οι κανόνες θα ισχύουν και για τον δημόσιο τομέα και για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι προφανώς ότι υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στον δημόσιο τομέα και γι' αυτό ακριβώς και έχω προτείνει ε, μια οδηγία έτσι ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ευελιξία και για τον δημόσιο τομέα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και οι συζητήσεις για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και οι συζητήσεις επίσης για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Νομίζω ότι μέσω των συζητήσεων αυτών θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο πάντα προστασίας για τους πολίτες να προωθήσουμε την ενιαία αγορά και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Μία επιπλέον φράση για το γιατί έχουμε εμείς επιλέξει τη μέθοδο της οδηγίας. Να προσθέσω εδώ και ακόμα και αν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία από πλευράς κρατών μελών την οδηγία την σχετική με τα θέματα ασφαλείας, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν εδώ συγκεκριμένες ρήτρες προστασίας. Οι κανόνες και τα δικαιώματα τα οποία εφαρμόζονται και στα δύο επίπεδα θα πρέπει να είναι ταυτόσιμοι. Αν το συγκρίνει αυτό κανείς με την απόφαση πλαίσιο την οποία έχουμε μπροστά μας, η οδηγία είναι ένα επιπλέον βήμα θα έλεγα, γιατί όχι μόνο καλύπτει τα θέματα της διαμεθοριακής συνεργασίας, αλλά καλύπτει επίσης και τις εσωτερικές διαργασίες, τις εθνικές διαργασίες από τις υπεύθυνε αρχές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχει κάνει και στα πλαίσια της απόφασης για τη υιοθέτηση ε, της πρότασης για την απόφαση πλαίσιο. Αυτά είναι θέματα λοιπόν και συμφώνησα και με τον κύριο Δρούτσα ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις αλλά επαναλαμβάνω ότι ε, στόχος είναι και οι δύο αυτές προτάσεις και οι δύο αυτές πράξεις να διευκολύνουν τα πράγματα, να δημιουργήσουν υψηλά επίπεδα προστασίας και να παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περιμένω με ενδιαφέρον λοιπόν τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν στις 8 και 9 Οκτωβρίου στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής συνάντησης του Κοινοβουλίου, δηλαδή με τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έχει καταστήσει τη συνάντηση του μηνός Οκτωβρίου εφικτή τα συγκεκριμένα επιμέρους έγγραφα εργασίας και οι προτάσεις εκθέσεως, εκθέσεων του κυρίου Δρούτσα και του κυρίου Άλμπερτ θα είναι δύο σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει όλη την φροντίδα η οποία χρειάζεται και σε επίπεδο της Προεδρίας και σε επίπεδο εργασίας κοινοβουλευτικής. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Κυρία Ρέντινγκ, μας κάνατε μια πάρα πολύ αναλυτική παρουσίαση των βασικών συστατικών του προγράμματος εργασίας σας. Αναφερθήκατε στις προτεραιότητες που υπάρχουν στον τομέα της δικαιοσύνης σε τρία βασικά θέματα. Πρώτον, την προοπτική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, το πακέτο ε, δικαστικής συνεργασίας, τα διαδικαστικά δικαιώματα και τρίτον, προστασία των δεδομένων. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί στη συνεδριάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επανειλημμένα και μάλιστα πολύ πρόσφατα, χτες όπως είπατε και ενεπλάξαν στη συζήτηση και οι δύο εισηγητέ και για τον κανονισμό και για την οδηγία. Για να υπάρξει λοιπόν μια τάξη στη διαδικασία θα ήθελα να πάρουμε μια πρώτη σειρά ερωτήσεων που να έχουν σχέση με το πρώτο θέμα, την πρωτοβουλία δηλαδή για τον διακανονισμό και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μέσω ποινικών μέσων. Και μετά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων, ο οποίος αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα και μετά ένας τρίτος γύρος ερωτήσεων σχετικά με, τα, με την προστασία των δεδομένων. Έτσι θα προστατευτούμε από το να, να αναμίξουμε τα θέματα και θα καταστήσουμε ικανή και την κυρία Ρέντινγκ να είναι παρούσα και να δώσει απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις τις οποίες θα θέσετε. Η κυρία Ρέντινγκ μου μίλησε με πολύ άμεσο τρόπο με διασφάλισε για τη συνεργασία της με την Επιτροπή στον συγκεκριμένο τομέα, στους συγκεκριμένους τομείς καλύτερα. Και γι' αυτό οφείλω και εγώ έτσι, να κάνω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η Επιτροπή μας και το Προεδρείο της Επιτροπής να έχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, να διασφαλίσει τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να είναι δραστήριο στον διοργανικό διάλογο και σε σχέση με τον διάλογο με, τις, με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Η συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου και σχετικά τώρα με την πρόταση για οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είμαι απολύτως πεπισμένος για την ανάγκη ε, να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα. Δεύτερον, Έχω σημειώσει δυστυχώς ότι λόγω των τεραστίων διαστάσεων της δημοσιονομικής κρίσης η οποία χαρακτηρίζει και σοβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όλες αυτές οι φιλόδοξες πλευρές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν αρχίσει να αγνοούνται θα έλεγα εν πολύ σε επίπεδο πολιτικής συζήτησης Ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα είναι ότι οι διαστάσεις αυτές συνδέονται, η οικονομική κρίση υπογραμμίζει τη σημασία για να υπάρξει πρόοδος στον τομέα αυτό, να έχουμε τα κατάλληλα μέσα και την βούληση να μπορέσουμε να αντιδράσουμε από κοινού εναντίον κάθε μορφών απειλών που θα υπονομεύσουν ακόμα περισσότερο την οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πράγματι το να έχουμε μπροστά μας έναν ορίζοντα μέσα στον οποίο να δουλέψουμε επί τη βάση του άρθρου 86 και να θέσουμε σε λειτουργία μια εμβριακή έστω μορφή ευρωπαϊκού εισαγγελέα, όχι μόνο για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακόμα και για τα εγκλήματα, ό,τι έχουν σχέση με το άρθρο 83, ακόμα και με την τρομοκρατία, με την σωματεμπορία, με την εκμετάλλευση των παιδιών, με το κυβερνοέγκλημα, με την ε, πορνογραφία στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι θέματα λοιπόν τα οποία καλείται ε, να αντιμετωπίσει ένας νομοθέτης Ευρωπαίος όπως είμαστε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα σαν παράδειγμα να γνωρίζω γιατί η οδηγία η σχετική με τη νομική βάση του άρθρου 125 και όχι με το άρθρο 83. Μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση εδώ έτσι ώστε η διαφθορά και η έκπληνση βρώμικου χρήματος που πραγματικά δημιουργούν απειλές ουσιαστικές στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Για μας λοιπόν αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, θα έλεγα, κάνοντας ένα πείραμα στον τομέα της ποινική ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε και θα δώσω τώρα το λόγο σε αυτούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος στη συζήτηση για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ευρωπαίος Εισαγγελέας και χρήση ποινικού δικαίου εναντίον απειλών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. The first hand that been raised, it's Mrs. Latford. We will be having a series of. Uh, Η κυρία Λάτφορντ αρχικά και μετά θα συνεχιστεί ο γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων από την κυρία Ρέντινγκ. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπω και εσεί. θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την ε, Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ που μας έκανε αυτή την ε, πολύ χρήσιμη ενημέρωση και μας δίνετε τη ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της κάποια ζητήματα σε βάθο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το προτινόμενο μέτρο για την καταπολέμηση της απάτης ε, κατά του προπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δράση σε αυτό το τομέα ε, Βεβαίω οι ευρωβουλευτέ συνεχώ ε, πρέπει να υπερασπίζονται αυτού ε, σε ερωτήματα του τύπου γιατί δεν κάνετε κάτι για την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί του προπολογισμού. Ω πολιτικοί λοιπόν ε, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα. Ε, με απασχολεί ιδιαίτερα η πρόταση για τις ελάχιστες κυρώσεις. Πριν από ένα χρόνο μόλις, και μάλιστα θυμήθηκα ότι ήταν ακριβώς στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή τότε λοιπόν ε, εξέδωσε ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και εμείς ε, ε, κάναμε, υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα φέτος και παραθέτω ενώ τα μέτρα ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμπληρώνουν τα εθνικά συστήματα ποινικού δικαίου, είναι σαφές ότι το ποινικό δίκαιο αντανακλά τις ε, βασικές ε, επιλογές και αρχές κάθε κοινωνίας και η συνθήκη της Λισαβόνας αποδέχεται αυτή την ποικιλομορφία. Εμείς στο δικό μας ψήφισμα, στο ενέκθεση De Jong τον Απρίλιο, υπογραμμίσαμε ότι οι προτάσεις για τέτοιες ουσιαστικές διατάξεις ποινικού δικαίου πρέπει να σέβονται απολύτως τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας. Όμως ε, αυτό που κάνουμε πάντα στις κυρώσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι τα δύο άκρα, μέγιστες και ελάχιστες. Όμως εσείς ε, διατίθεστε να υπάρχει και διακριτική ευχέρεια, δηλαδή με κάποια κριτήρια ο δικαστής θα πρέπει, συγγνώμη αλλά υπάρχει αρκετή φασαρία και αποσυγκεντρώνομαι. Ο δικαστής λοιπόν θα πρέπει να καταδικάζει κάποιον σε τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση. Εγώ προτείνω, Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ, ε, θεωρώ μάλλον ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ε, προϋπόθεση αναλογικότητας ε, στις κυρώσεις που εγγράφονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και έτσι μπορούμε να φτάσουμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια λόγω τέτοιας διάταξης. Επομένως, υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση στις αρχές της αναλογικότητας και περικορικότητας δεν ξέρω τα νομικά συστήματα άλλων χωρών, αλλά σίγουρα στη δική μου η διακριτική ευχέρεια των δικαστών είναι ε, θεμελιώδη σημασία ε, στοιχείο του, του δικαστικού μα ζητήματο. Βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ ότι κάποιο δικαστή πρέπει να ε, βγάλει μια καταδίκη, μια κύρωση, όσο δυσανάλογη και αν είναι η ποινή. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ισόβια κάθριξη χωρί δυνατότητα αναστολή. ο πρόεδρος ε, είναι μάλλον λίγο ανυπόμονος, μόνος τελειώνω, ε, να πω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο ε, μπροστά σε επόμενα μέτρα. Θεωρώ ότι είναι λάθος η προσέγγιση. Πρέπει να μείνουμε σε αυτή την αρχή του, των αλλάγιστων και μέγιστων ποινών και να αφήσουμε ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ε, δικαστικής. Okay, thank Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα τώρα είναι ποιος θέλει να υποβάλει ερωτήματα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Είπατε και για τον εισαγγελέα. Ναι, βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος, γιατί κινείται στην ίδια λογική. Κυρία Σίπελ και μετά κυρία Σαρτζεντίνη. Uh, Θα κάνουμε τρεις γύρους ερωτήσεων για να μπορεί και η κυρία Ρέντινγκ να σας απαντήσει λίγο πιο δομημένα. Ο πρώτο γύρο ερωτήσεων αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τον εισαγγελέα. Μετά δικονομικά δικαιώματα και μετά προστασία δεδομένων. Πρώτο γύρος ερωτήσεων λοιπόν, κυρία Σίπελ. Εκτό μικροφώνου. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα, αλλά θα ήθελα να σα πω ότι θέλω και στα άλλα δύο σημεία να θέσω κάποιο ερώτημα. Για τα, χρηματο... για τα χρηματικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορώ να είμαι σύντομη. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω δεν χρειαζόμαστε οδηγία για να το λύσουμε. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται κάπου στα κράτη-μέλη και γι' αυτό θέτω το ερώτημα και αυτό είναι και το ερώτημα που απευθύνω στην κυρία Ρέντινγκ πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας όταν ήδη στα κράτη-μέλη εκεί πάλι πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία κατά της απάτης εναντίον του προϋπολογισμού. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, αποφασίζουμε κάτι το οποίο είναι γενικό, αλλά μετά το πώς εφαρμόζεται αυτό, πόσο αποτελεσματικό θα είναι, δεν το ξέρουμε. Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. άκουσα τις προτάσεις για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και γύρονται κάποια ερωτήματα. Προχωρούμε προς την δικαστική συνεργασία. Ε, μια μορφή αυτής της συνεργασίας είναι και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, όμως ε, αφήνουμε εκτός ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η σαφές ε, πολιτική, σαφής πολιτική για την ε, νομική αρρωγή. Αν υπάρχει ε, εισαγγελέα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και θα έχουν την κατάλληλη νομική αρρωγή οι πολίτες. πολλά λέγονται για την πρόσβαση σε δικηγόρο, αλλά στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει νομική αρρωγή, σε άλλα όχι. Και αν κάποιο δεν έχει νομική αρρωγή, η πρόσβαση σε δικηγόρο μάλλον δεν ισχύει. Χθες ε, ψηφίσαμε επί της ε, οδηγίας ε, για το Δουβλίνο και για τους ετούντες άσυλο. Σε αυτά τα κείμενα αναφέρεται και πάλι νομική αρρωγή. Όμως αν δεν προβλέπεται νομική αρρωγή σε ένα κράτος μέλος, τότε πώς μπορεί ο ο ετών άσυλο να λαμβάνει τέτοια νομική αρρωγή, ενώ ο πολίτης όχι. αναφερθήκατε στους ευάλωτους υπόπτους υπάρχει μια πρόταση, δεν είμαι σίγουρη, αλλά και πάλι, αν οι ευάλωτοι, οι ύποπτοι πράγματι χρειάζονται νομική αρρωγή, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δεν ε, προβλέπει υποχρέωση ύπαρξης ε, συνηγόρου και στις δύο πλευρές. Σας έχω πει 15 φορές ε, έχω αναφέρει τον όρο νομική αρρωγή, αλλά θεωρώ ότι αν θέλουμε να εργαστούμε επί της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την παροχή νομικής αρρωγής στους πολίτες. Και άκουσα ότι δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει τέτοια πρόταση μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ε, διερωτώ με λοιπόν αυτό ισχύει και αν ναι, αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί για να μπορέσουμε πραγματικά να πιστέψουμε στη δικαστική συνεργασία στην Ευρώπη και για να πούμε στους πολίτες μας ότι θα προστατευθούν ε, έναντι μιας απόφασης ε, ε μάλλον ερεύνη από άλλο κρατό μέλο, πρέπει να υπάρχουν κάποια εχέγγυα. Αυτό είναι το ερώτημά μου λοιπόν προ εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταπολέμηση του διασυνοριακού ε, εγκλήματος και τη τρομοκρατία, όλα αυτά απαιτούν ε, ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία στα ζητήματα ποινικού δικαίου. Και εδώ φτάνω στο ζήτημα της εμπιστοσύνης που είναι ουσιώδης σημασία για την ε, δικαστική συνεργασία και για να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμα δικονομικά συστήματα. Επομένω, ε, σκέφτεστε να, να προτείνετε έναν τρόπο αξιολόγηση ε, των δικαστικών αυτών ζητημάτων, ε, συστημάτων στα κράτη-μέλη, να δούμε πού υπάρχουν οι βέλτιστε πρακτικέ, να τι υλοποιήσουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Ιδάλω, αν δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των συστημάτων, δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη και έτσι δεν, μπορεί, ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ταχεία και αποτελεσματική δικαστική συνεργασία και η ανταπόκρισή μας ε, στην τρομοκρατία και στο οργανωμένο έγκλημα δεν θα είναι ε, η χρηστή. Ευχαριστώ. Κυρία Μπατιέ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Είναι καλά νέα αυτά που μας φέρνει η κυρία Ρέντιν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσχεση του, των στοιχείων ενεργητικού των ε, εγκληματιών, για την εισαγγελική αρχή για τα θέματα αυτά. Για το τελευταίο βέβαια θα ήθελα κυρία Ρέντινγκ να μας πείτε λίγο περισσότερο παρά το γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και για τη Κομισιό και για τα κράτη-μέλη και για ορισμένες πολιτικές ομάδες. Εγώ συμμερίζομαι λίγα και την άποψη του Πρόεδρου. Γιατί από τη στιγμή που η Κομισιόν εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ε, εισαγγελικής αρχής, γιατί να περιοριστεί αυτή η αρχή μονάχα σε ένα στενό τομέα. Εγώ νομίζω θα έπρεπε να καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο. Έχουμε μιλήσει παραγωγικά για θέματα όπως είναι η παιδοφιλία και άλλα θέματα εγκληματικότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή την αρχή, γιατί να μην καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων. Χαιρετίζω εξάλλου τι ε, πρωτοβουλίε τη Κομισιόν προ την κατεύθυνση αυτή. Το Κοινοβούλιο, όπω ξέρετε, έχει δημιουργήσει μια επιτροπή, μια έκτακτη επιτροπή, την Επιτροπή Κρίμη, με πολλά μέλη τη Επιτροπή Λίμπη που είναι σήμερα παρόντα. Έχει ακούσει τι ε, παρεμβάσει συνομιλητών όπω είναι η Ευρωζήστ, η Ευρωπόλ, τα μέλη τη Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν ένα ιδιαίτερα έφορο χώρο ο οποίο είναι ανοιχτό στου ε, εγκληματίε λόγω τη ε, οικονομική κρίση. Η μαφία βρίσκει λοιπόν αυτό το έφορο έδαφο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τη και επομένω οποιαδήποτε προσπάθεια τη Κομισιόν κατά του οργανωμένου εγκλήματο είναι ιδιαίτερα καλόδεκτη από εμά. Βοργέτσιο. Πιάνομαι από την τελευταία παρέμβαση για να επιμείνω κι εγώ σαν Ιταλός βουλευτής να επιμείνω ζητώντας την προσοχή σας, Επίτροπε. Σας συγχαίρω κατά τα άλλα βέβαια για την αποφασιστικότητα η οποία σας χαρακτηρίζει στην περίπτωση αυτή της πρότασης οδηγίας, ειδικά σε σχέση με την ανακύκλωση χρημάτων και ε, τις απάτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και για τις εργασίες της δικής μας της ειδική Επιτροπής ΚΡΙΜ θα πρέπει η Επιτροπή να μας ενημερώσει όσο καλύτερα γίνεται. Επιμένω λοιπόν για το θέμα της συμμετοχής των εγκληματικών τύπου οργανώσεων όπως η μαφία σε τέτοιου δραστηριότητες. Εγώ ήμουν μέλος σε μια παλιά επιτροπή εναντίον της μαφίας στη χώρα μου και τότε συζητούσαμε ε, για τις κοινοτικέ απάτες, τη συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος και την ανάγκη να αντιπαρατεθούμε με αυτό. Εν πάση περιπτώσει το θέμα τίθεται πάντα και είμαι βέβαιος ότι τεκμήρια υπάρχουν πάρα πολλά ήδη διαθέσιμα. Τηλεγραφικά ένα άλλο ερώτημα εδώ, ιδιαίτερα επίκαιρο. Πιστεύετε άραγε η κυρία Ρέντεν και πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα ότι μιας και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία και σε όλες τις διπλωματικές αποστολές της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά από την δημοσίευση στο σατυρικό εβδομαδιαίο περιοδικό Σαρλί Hebdo. Στην ουσία αύριο κλείνουν όλες τις διπλωματικές τους αντιπροσωπείες. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια αφορά άμεσα τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αλλά θα πρέπει να επαναλάβουμε το άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας και την εμβέλεια της Χάρτας των Δικαιωμάτων έτσι ώστε να διασώσουμε θα έλεγα την νομική αρχή της ελευθερίας ε, έκφρασης και της ελευθερίας σάτυρας που είναι ένα από τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού και φυσικά αυτό το θεμέλιο θα πρέπει να το σεβαστούμε σεβόμενοι βέβαια τις ευαισθησίες αυτών οι οποίοι νιώθουν ότι προσβάλλονται. Σε άλλες περιπτώσεις όταν πρόκειται για ένα θα έλεγα ένα φίλμα παράδεκτο, προσβλητικό κτλ. Αυτό είναι καταδικαστέο. Αλλά εγώ αναφέρομαι στη σάτυρα. Και το ότι οι hacker χθε μπλόκαραν την ιστοσελίδα του περιοδικού αυτού, δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει, δεν μπορούσε να στείλει φάξ. Και προσπάθησα και εγώ να έρθω σε επαφή μαζί με το Σαβλί Εμπτό. Αυτό είναι σκάνδαλο για την Ευρώπη των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέντινγκ, αυτά τα οποία λέτε ακούγονται πολύ καλά. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα υπάρχουν ελλείμματα εκεί. Μιλήσατε για 600 εκατομμύρια τα οποία χάνονται, τουλάχιστον. Αυτό λοιπόν το κατανοώ. Από την άλλη πλευρά όμως έχω κάποιο σκεπτικισμό. Όχι για τον στόχο τον οποίο θέλετε να επιτύχετε, αλλά για, τον, για τις δυνατότητες κυρώσεων θα πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι τα κολάσιμα δικήματα, πώς θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η απάτη φαίνεται ότι είναι ένα απλό θέμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια σαφήνεια σε σχέση με τους ορισμούς στον τομέα αυτό. Δεν ξέρω αν ο δρόμος που προτείνεται είναι ο καλύτερος. Είμαι έτοιμη να με πείσετε όταν μιλάτε για Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Εγώ δεν κατανοώ αυτό ότι για ένα συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εισαγγελική αρχή. Τι γίνεται με το εθνικό δίκαιο, πώς συνάδει αυτό με το εθνικό δίκαιο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε ένα περιορισμένο πεδίο μπορεί να υπάρχει μια υπερεθνική ευρωπαϊκή αρχή. Και τίθεται φυσικά και το θέμα της εναρμόνισης σε ό,τι αφορά την ε, δικαιοσύνη. Εν γέννη, βλέπετε <clears throat> να υπάρχουν βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με την κατεύθυνση των κρατών μελών προς μια εναρμόνιση. Είναι πρόθυμα τα κράτη να προχωρήσουν προς μια α, εναρμόνιση ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μελλοντικό εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακιντάρ θέλει και αυτή να λάβει Μόνο να θίξω ένα ζήτημα σε σχέση με, τον Ευρωπαϊκό, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Εγώ βλέπω να υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης με το έργο το οποίο γίνεται ήδη από τα κάτι μέρη. Σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα να υπάρξει επικάλυψη με το έργο της Ευρωζούστου. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα τη συνεργασία, τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών. <clears throat> Αλλά έχω ανησυχίες και κατά πόσο η δημιουργία νέων πολυδάπανων φορέων θα μπορέσει να οδηγήσει σε πραγματική προσθεμένη αξία η σειρά σας τώρα κυρία Επίτροπε Ρέντινγκ να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων για να περάσουμε στα επόμενα σημεία μετά. Να ξεκινήσουμε με την εισαγγελική αρχή. Γιατί να δημιουργήσουμε σε ένα τόσο περιορισμένο πεδίο δράσης. Γιατί να μην επεκτείνουμε την αρμοδιότητα αυτής της αρχής, αρχής γενικά στα διαμεθοριακά αδικήματα. Καταρχήν υπάρχει ένα πρόσκομα από τις συνθήκες. Οι συνθήκες με τρόπο σαφή και νομίζω απόλυτα αιτιολογημένο περιορίζουν τις δυνατότητες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό με συνδέει κατευθείαν στο ερώτημα, με το ερώτημα της κυρίας της Βαρόνης, Λατφόρτ. Γιατί η συνθήκη <clears throat> δεν προχωράει περισσότερο στα θέματα αυτά. Γιατί η ποινική δικαιοσύνη είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας, ο οποίος συνδέεται με την αρχή της επικορικότητας και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας είπα και το επαναλαμβάνω και παραμένω και επιμένω στο σημείο αυτό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το πώς επιζητούμε την εναρμόνιση στον τομέα της ποινική δικαιοσύνη. Προς το παρόν, η συνθήκη λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε ζητήματα που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τις πολιετής προοπτικές. Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε πέραν αυτού, τότε είναι απαραίτητη μια αλλαγή των συνδικών. Αυτό είναι εύλογο, αν σκεφτείτε το πρόβλημα του διαμεθοριακού εγκλήματος και ο πρόεδρος ανέφερε και άλλα, άλλους χώρους όπου υπάρχουν νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαμεθοριακό έγκλημα. Για να μπορέσουμε όμως να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, δεν μπορούμε προς το παρόν να το πράξουμε επί τη βάση της συνθήκης ως έχει. Εγώ υποστηρίζω την αλλαγή της συνθήκης. Αλλά στην περίπτωση αυτή, προς το παρόν και είναι ορθό και πρέπον, είμαστε υποχρεμένοι να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση βήμα-βήμα και να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία μας επιτρέπει να πράξουμε συνθήκη. Ο πρόεδρος επίσης, ο πρόεδρος έθεσε το ερώτημα αυτό της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί διαλέξαμε σαν νομική βάση για το τρομοθέτημα αυτό το άρθρο, το άρθρο 325 και όχι το άρθρο 83 για να το θέσω με απλά λόγια. Γιατί το άρθρο 325 καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε να φανταστείτε. Και συγγνώμη και ο λόγος για τον οποίο παρεμβαίνουμε είναι γιατί εδώ δεν έχουμε μία επίθεση, μία ζημία προς, τον, προς ένα εθνικό προϋπολογισμό αλλά αντίθετα μια ζημία, μια επίθεση κατά του κοινού μας ταμείου του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Μπορείτε να φανταστείτε να μην αντιμετωπίσουμε τους εγκληματίες σε κάποια κράτη-μέλη. Να υπάρχει εξαίρεση σε, για τους εγκληματίες ορισμένων κρατών μέλων όταν προβαίνουν σε απάτες ή άλλες επιθέσεις κατά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα προέκυπτε, αν είχαμε μια διαφορετική νομική βάση, γιατί τότε μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα της αυτοεξαίρεσης, του opt-out από ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν θα ήταν ο ορθός τρόπος να προχωρήσουμε, γιατί και πάλι θα οδηγούσε σε εμβαλωματικές λύσεις και τη δυνατότητα των εγκληματιών να υπεκφεύγουν. Το άρθρο 325 αναφέρεται σε μέτρα τα οποία, παραθέτω, θα μπορούσαν να δράσουν ως αποτρεπτικά στοιχεία πέρας της παράθεσης. Η διατύπωση αυτή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο σοβαρών αδικημάτων απάτης και αυτό καταδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το άρθρο ως η βάση για μέτρα στο ποινικό δίκαιο <clears throat> και αν δείτε πως έχει εξελιχθεί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προηγούμενο άρθρο στον τομέα αυτό εκπεφρασμένα απέκλειε μέτρα τα οποία έχουν επίπτωση στην εφαρμογή της εθνικής, του εθνικού ποινικού δικαίου. Αυτό όμως ήταν πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα το τωρινό άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν εκ... αποκλείει πλέον την εφαρμογή την ε, εφαρμογή του εθνικού ποινικού δικαίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μέτρα εθνικού ποινικού δικαίου και όπως είπα προηγουμένως απαντώντας στον πρόεδρό σας, είναι πολύ σημαντικό όλα τα κρατη να συμπεριληφθούν σε μια τέτοια πρόνοια γιατί δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τις απάτες και τις ζημίες προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα διαμεθοριακά δικήματα. Είναι απειλές και επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως θα πρέπει τα μέτρα εναντίον τους να ισχύουν σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The question... Τώρα, για το θέμα του πώς τα κάτι μελη θα ενσωματώσουν στην ένωμη τους, στην εθνική ένωμη τάξη αυτή την οδηγία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντα αντιμετωπίζουμε με οποιοδήποτε νομοθέτημα που έχει τη μορφή οδηγίας. Πάντα είναι θέμα του πώς θα μεταγραφεί αυτή η οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Κομισιόν φυσικά συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη κατά την διάρκεια της διαδικασίας μεταγραφής. Και είναι σαφές ότι ο, η Κομισιόν ως θεματοφύλακας των συνθήκων, εάν θεωρήσει ότι η μεταγραφή δεν έχει γίνει με τρόπο σύμμορφο με την οδηγία, μπορεί πάντα να παρέμβει και να προσφύγει σε τελική ανάλυση και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι θέλετε να διαχωρίσετε τα διάφορα επιμέρους ερωτήματα. τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν δείχνουν ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός σε κουτάκια. Γιατί συνδέονται μεταξύ τους τα θέματα αυτά. Και η κυρία Σαρτζεντίνη έθεσε το ερώτημα της νομικής αρρωγής και γιατί δεν έχουμε, και του γιατί δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει το θέμα της νομικής αρρωγής στην οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο ερώτημά της. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σαρτζεντίνη ότι είναι θεμελιώδες στοιχείο προς την κατεύθυνση μιας δίκαιας δίκης η νομική αρρωγή. Το αναφέρει και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και η οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο <clears throat> πάντα αντιμετώπιζε τα ουσιαστικά δικαιώματα σε σχέση με πρόσβαση σε δικηγόρο. Το θέμα της νομικής αρρωγής όμως είναι πιο πολύπλοκο και χρειάζεται μια πιο λεπτομεριακή ανάλυση αντικτύπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πέσει σε μια μαύρη τρύπα, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κανόνων για τη νομική αρρωγή το δικαίωμα για νομική αρρωγή προνοείται στο άρθρο 6 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο άρθρο 7 της ε, ίδιας Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλα τα κρατη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να υλοποιήσουν ένα αποτελεσματικό, αποτελεσματικά το δικαίωμα στη νομική αρρωγή χωρίς διάκριση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών σε ορισμένες περιπτώσεις. <clears throat> Επί, επειδή όμως κατά τη διάρκεια της ανάλυσης που κάναμε είδαμε ότι αυτό το στοιχείο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη σε μία δήλωση του Συμβουλίου τον Ιούνιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εγώ δεσμεύτηκα να προβώ και σε μία ανακοίνωση για την νομική αρρωγή, ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος κανόνας για τα θέματα αυτά. Παραμένει πάρα πολύ πολύπλοκη κατάσταση, υπάρχουν μεγάλες πολυπικιλίες ρυθμίσεις ως τα κράτη-μέλη, γι' αυτό προτού μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική έκθεση αντικτύπου, θα πρέπει να έχουμε προηγουμένως μια λεπτομερή μελέτη συγκριτικού χαρακτήρα η οποία μετά μπορεί να είναι η βάση για την πρόταση νομοθετικών μέτρων στον τομέα αυτό. Αυτή η μελέτη είναι αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία. Εξετάζουμε λοιπόν και εργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Αυτό με τη σειρά του συνδέεται με το άλλο ερώτημα της εμπιστοσύνης. Το σύστημά μας δεν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει τους ε, εθνικούς ε, νόμους και κανόνες. Ε, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ελάχιστα δικαιώματα και κανόνες και να γεφυρώσει τα χάσματα μεταξύ των επιμέρους συστημάτων. Αυτό το βασικό στοιχείο για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα είναι η εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δεν λειτουργεί το σύστημα. Το είδαμε τώρα αυτό με το ένταλμα σύλληψης, όπου οι δικαστές αποφασίζουν να μην ε, το, εφαρμόσουν, να μην το εκτελέσουν, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους ε, νόμους ε, των γειτονικών κρατών μελών. Είναι σαφές λοιπόν ότι όλο το σύστημα της εμπιστοσύνης είναι ζωτική σημασίας ε, για το εγχείρημα αυτό. Γι' αυτό και είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα παρακολούθησης των δικαστικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρακολουθούμε για την οικονομική ανάπτυξη στοιχεία της, ε, στοιχεία της οικονομικής ζωής αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της ε, διοίκησης. Ενώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ε, χώρες ε, που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα, τις βοηθάμε λοιπόν να ε, διαμορφώσουν και να χτίσουν ένα υγιές σύστημα, είδαμε ότι υπάρχει ε, άμεση σύνδεση μεταξύ της μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας των ε, αστικών, εμπορικών και ποινικών συστημάτων και της, και της διστακτικότητας για επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Και εκεί διαμορφώθηκε και γεννήθηκε αυτή η ιδέα ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην έχουμε μόνο στοιχεία που συνδέονται ξεκάθαρα με την οικονομία και την κοινωνία, αλλά να συμπεριλάβουμε και στοιχεία που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Προς το παρόν, πέρα από τους ε, αρμόδιους πραγματογνώμονες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Έχουμε θέσει επιτάπητος ε, τα κάποια στοιχεία προκειμένου ε, σε αυτές τις χώρες να υπάρχουν συγκεκριμένες αναλύσεις και συστάσεις, ειδικέ συστάσεις για την αναθεώρηση, αναδιάρθρωση του συστήματος ε, δικαιοσύνης σε αστικά και εμπορικά ζητήματα ανακοίνωσα για την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο ότι θα υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το ανακοίνωσα και στους υπουργού χθες το απόγευμα στη Βιέννη, όπου έγινε συνάντηση των 27 υπουργών και των 27 ε, μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τους υπουργούς δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από αυτό που εγώ αποκαλώ δίλημα της Κοπεχάγης. Αφενός έχουμε χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν. Ε, τις ε, παρακολουθούμε ε, στενά και τις ε, πιέζουμε, τις βοηθάμε να, να οικοδομήσουν ένα τέτοιο σύστημα Έχουμε πάσει πάνω τους λοιπόν και όταν αυτές οι χώρες ε, γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η δυνατότητα παρέμβασής μας είναι πολύ περιορισμένη. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάση και το άρθρο 7, ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέτρα δεν υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο εργαλείο. Και έτσι η περαιτέρω διαμόρφωση αυτού του βαθμολογίου για την δικαιοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά πρέπει πρώτα να επιληθεί ε, το δίλημα αυτό. Με ρωτήσατε για την ε, εισαγγελική αρχή και μήπως έτσι υπάρχει επικάλυψη του έργου της Eurojust. Η Eurojust είναι ένας μάλλον χαλαρός οργανισμός ε, όπου ε, οι εισαγγελείς των κρατών μελών συναντιούνται ξεκίνησε ως μια προσπάθεια στενότερης συνεργασίας. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι σε ζητήματα που συνδέονται με το έγκλημα κατά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο, η Εθνική Εισαγγελική Αρχή σταματά στα σύνορα του κράτους μέλους. Και αν στο παραδίπλα κράτος μέλος δεν υπάρχουν κανόνες και δεν θεωρείται κάτι τέτοιο αξιόπινη πράξη, βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να ορίσουμε το έγκλημα και τις ε, ελάχιστες χειρώσεις και μετά ε, να φέρουμε τους, τις εγγελικές αρχές σε στενότερη συνεργασία. Βεβαίως και αυτό είναι κάτι που ε, ε, συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα έγγραφα που έχει εξετάσει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ότι πρέπει δηλαδή να υπάρξει εξέλιξη ε, της Eurojust και να γίνει ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή βάσει των στοιχείων που προβλέπονται στην συνθήκη. Έτσι προχωρούμε λοιπόν βαθμιαία. Ε, δεν θέλω να κάνω ότι δεν άκουσα του κυρίου Μοργέτσιο, γιατί βεβαίως και μας αφορά ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Γι' αυτό και όλοι αυτή τη στιγμή αυτό συζητούν. Σε τι ακριβώς συνίσταται το δικαίωμα της ελευθερίας και το δικαίωμα στη σάτυρα που συνδέεται με την ελευθερία έκφρασης. Βεβαίως και αυτή η αρχή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατίας μας. Και γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο σε τέτοιες ε, περιπτώσεις να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία. Εγώ ως ε, πρώην δημοσιογράφος έχω ένα στοιχείο πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι η ελευθερία έκφρασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατίας μας. Ευχαριστώ Επίτροπε. Λοιπόν, προβλέπετε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά α, μέχρι τις 5 γιατί μετά έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα δυστυχώς τα οποία είναι σχετικά. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Έχω τουλάχιστον 10 μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Δώδεκα μέλη έχουν ζητήσει το λόγο, όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Έτσι ώστε η Επίτροπος να έχει χρόνο να απαντήσει για τα θέματα των διαδικαστικών δικαιωμάτων και για την παρακράτηση των δεδομένων. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δρούτσα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα, εισηγητής. 15 δευτερόλεπτα να κάνω μια παρατήρηση. Εκτός από τα τρία θέματα τα οποία επιλέξατε, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να θέσουμε σήμερα. Και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλο είναι το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ρέντινγκ και γι' αυτό μέχρι τις 5 να σκεφτείτε παρακαλώ για το πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Κοιτάξτε, από εσά εξαρτάται. Στον πρώτο γύρο υπήρξαν πολύ περισσότερες ερωτήσεις και όχι μόνο για τα οικονομικά συμφέροντα ή για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε λοιπόν σε αυτό το γύρο την προσοχή σας στα θέματα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να τεθούν για τη συζήτηση. Ο κύριος Βρούτσας πάντως έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος και θα ασχοληθώ με το θέμα των ε, προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Να δηλώσω ότι έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την Επίτροπο Ρέντινγκ και τις υπηρεσίες της. Εξαιρετική συνεργασία. Να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ρέντινγκ για το φιλόδοξο πλαίσιο το οποίο έχουμε. Εμένουμε μεν αλλά από την άλλη θεωρούμε ότι η ποιότητα προηγείται και αυτή είναι η δύσκολη ισορροπία την οποία πρέπει να κρατήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να στραφώ τώρα στο θέμα της οδηγίας. Όπως είπατε και εσείς, κάνατε συγκεκριμένες ε, επιλογές στην πρώτη φάση, ένα κανονισμό και τα οδηγία κτλ. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προτιμούσαμε να είχαμε ένα νομικό μέσο ένα νομικό κανονισμό που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων προστασίας δεδομένων. Παρ' όλα αυτά δεχόμεθα και ε, τις επιλογές τις οποίες κάνατε. Εμείς βλέπουμε το θέμα αυτό της προστασίας των δεδομένων σαν ένα πακέτο. Σε αυτή τη συνολική αντιμετώπιση θα εμείνουμε και αν είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα, την, θα υπερασπιστεί τον χαρακτήρα αυτό που ε, είπα. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε κάποια ανησυχητικά μηνύματα από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου ότι ορισμένα από αυτά δεν θέλουν να προχωρήσουν με τη συγκεκριμένη οδηγία. Θα ήθελα να μας πείτε παρακαλώ αν έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των διαπραγματεύσεων στο εσωτερικό του Συμβουλίου για το θέμα που με ενδιαφέρει. Ποιες είναι οι ανησυχίες των κρατών μελών και ποια είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περίπτωση κατά την οποία τα νέα από εκεί δεν είναι πολύ ευνοϊκά. Ένα δεύτερο θέμα αφορά τον κανονισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο θέμα και πάρα πολλά είναι τα επιμέρους θέματα, οι συνάδελφοι θα αναφερθούν άλλωστε σε αυτά. Ένα να, με απασχολήσει, να σας απασχολήσει σε αυτή τη φάση η κατεξουσιοδότηση πράξης. Γνωρίζετε ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θεωρούμε την τεκμηρίωση την οποία παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το συνολικό αυτό το θέμα αν πράγματι χρειάζονται οι κατεξουσιοδότηση πράξεις ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχουμε κάποιες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε αυτό το νομοθετικό κενό με ένα νέο μηχανισμό ο οποίος θα καλύπτει ιδιαίτερα τα θέματα που θέτει η τεχνολογική πρόοδος. Κυρία Γκάλ, αναφερθήκατε προηγουμένως. Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Θεωρείτε ότι αν υπάρξει μία απόφαση ανωτά του δικαστηρίου σε εθνικό επίπεδο που αρνείται να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης θα μπορούσε να υπάρξει θεραπεία με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νομίζω ότι γνωρίζετε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και φαντάζομαι ότι το έχετε στο μυαλό σας όταν συζητάμε τα θέματα αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το δίλημα της Κοπενχάγης που αναφέρατε και το πίνακα επιδόσεων για τη δικαιοσύνη. Στα κριτήρια της Κοπενχάγης υπάρχει η απέτηση να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων. Αν είχαμε τώρα για τα θέματα αυτά ένα πίνακα επιδόσεων, το θέμα αυτό το οποίο φεύγει από τα χέρια της Κομισιόν όταν ένα κράτος μέρος προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και πάλι, γιατί τότε τουλάχιστον θα εμφανιζόταν σε αυτόν τον πίνακα επιδότηση ως κάτι το οποίο χρειάζεται πραγματικά με τα φαινόμενα που βλέπουμε. Κύριε Γκυγιόμ. Κύριε ε, Πρόεδρε, θα δώσω συνέχεια σε ορισμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Εγώ, αν θέλετε, εμπίπτω στον τέταρτο γύρο ερωτήσεων και αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να θίξω αυτά τα θέματα. Λοιπόν, παίρνω το λόγο. Τώρα, τώρα, κάντε το τώρα, λέω ο πρόεδρος. Θα μιλήσω, επομένως, για ένα θέμα διαφορετικό. Για τους Ρωμά. <clears throat> Επανέρχομαι λοιπόν για σε ένα θέμα. Για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχει τρεις πτυχές για μένα. Είναι θέμα της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής δράσης που θέλουμε να την, να δούμε να ενισχύεται. Το θέμα της, εφαρ... της ε, απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που δεν είναι πάρα πολύ καλό και εξακολουθούν να με ερωτήματα για το θέμα αυτό. Ήθελα να ξέρω αν έναντι των, ε, των ε, κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς λόγω προβλημάτων διοικητικών ή όχι. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το σημαντικό θέμα απορρόφηση κονδυλίων και πώς θα εξασφαλίσετε καλύτερη εκτέλεση αυτών των κονδυλίων. Δεύτερο ερώτημα. Οι εθνικές στρατηγικέ ενσωμάτωση δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Έχετε στα χέρια σα αυτέ τι στρατηγικέ και κάποιε από αυτέ ήταν και εκτό θέματο θα μπορούσα να πω. Θα ήθελα να ξέρω αν θα κάνετε κάτι για να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και δεν ξέρω πώς θα αξιολογήσετε την πρόοδο ή μη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των Ρωμά. Και τέλος το ερώτημά μου είναι αν σκέφτεστε να έχετε κάποιους, κάποιες νέους οδούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για προγράμματα παραγωγής χάρη οικονομικής επανενσωμάτωσης. Και εδώ μιλήσατε για θέματα συνεργασίας και τη χρήση μικροπιστώσεων και καλύτερη ε, προετοιμασία υποδοχής των μεταναστών για να αποφευθεί η ενεργοποίηση κυκλωμάτων μαφιόζων που θα τους εκμεταλλευτούν και επίσης αν έχετε άλλα μέτρα για τον τομέα αυτό εκτός από τα κατασταλτικά. Κυρία Κέλλερ. Και για τους Ρωμά, θα ήθελα και εγώ για τους Ρωμά. Τώρα υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και, και Ρουμανίας για την ε, αποστολή στη Ρουμανία, την επιστροφή των Ρωμά στη Ρουμανία, θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν τα αποτελέσματα των επαφών σας με την ε, γαλλική κυβέρνηση, επίσης για το θέμα της ε, Ευρωπόλ, τα θέματα δεδομένων. Η Ευρωπόλ θέλουν να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να μοιράζονται δεδομένα με τρίτες χώρες, με ιδιωτικούς φορείς, να μπορούν επίσης να μοιράζονται και ευαίσθητα δεδομένα, να έχουν δυνατότητα να συνδυάσουν τράπεζες δεδομένων. Αυτό μου φαίνεται ότι αντιβαίνει με, με την οδηγία για την προστασία δεδομένων. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς το βλέπετε αυτό σε σχέση με την οδηγία για την προστασία δεδομένων και ποια είναι η άποψή σας για την ε, αναθεώρηση του πλαισίου της Ευρωπόλ. ο Σένσιου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, θέλω να σας θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ξέρω για την πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα εξασφαλίσει το κράτος δικαίου, όπως παρουσιάστηκε από την κυρία Επίτροπο στο Στρασβούργο. Διατηρείτε την πρότασή σας αυτή ή όχι. Στη συνέχεια, δεν έχουμε ίσως πολύ χρόνο σήμερα το απόγευμα και γι' αυτό θέλω να μιλήσω εν συντομία και εγώ για το θέμα των Ρωμά και να σας πω ότι η λύση της ενσωμάτωσης δεν έχει λειτουργήσει μέσα σε μεμονωμένα κράτη-μέλη, νομίζω ότι απαιτείται μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει μια πραγματική αντιμετώπιση για τις κοινότητες στο Ρωμά. Εγώ έχω κάνει μια μεγάλη μάχη για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και στις χώρες όπου ζουν τώρα οι Ρωμά και επίσης να λάβουμε υπόψη και τον εμπειρογνωμών για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι η πρότασή σας για την ενσωμάτωση των Ρωμά δεν μπορούν να στεφτούν από επιτυχία εάν δεν συνοδεύονται από μια πραγματική δράση στον τομέα αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη θέση που έχετε αναλάβει για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και την συμπερίληψή τους στον χώρο Σέγγεν. Εγώ κατανοώ τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στη δήλωσή σας. Πιστεύω όμως ότι μια τέτοια θέση μπορεί να, έχει, να εμπεριέχει κινδύνους. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες δεν έχω διασταυρώσει απόλυτα, αλλά εδώ έξω από το Κοινοβούλιο, στο Πάρκο Λεοπόλτ, υπάρχουν ξενόφοβες αφήσει που ζητούν από το βελγικό πληθυσμό να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Είναι λοιπόν μια επικίνδυνη θέση η οποία έχει αναλυφθεί. Μπορεί κανείς να δει κάπως ε, διαφορετική την δική σας στάση από τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η Κομισιόν επίσημα, σαν σύνολο, δεν ήταν ποτέ κατά της ε, συμπερίληψης Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο αυτό. Κυρία Στάνοκα. Κύριε Επίτροπε, Θα ήθελα να αναφερθώ στη δήλωσή σας την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο Μήπως μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες περί τίνος πρόκειται. Τι ακριβώς εννοείται γύρω από το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και σύν της άλλης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την εφαρμογή των υπαρχουσών προβλέψεων και να δούμε αν υπάρχουν εμπόδια για την σωστή εφαρμογή και τον σεβασμό στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κυρία Γκόντς, θα είμαι πολύ πειθαρχημένη, θα ήθελα να είμαι πειθαρχημένη και να περιμένω μέχρι τον τέταρτο γύρο, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι βιαζόμαστε. Δύο ερωτήσεις αυτό το στοχολόγιο ή ε, το πίνακα επιδόσεων. Είχε τεθεί το θέμα αυτό και στα πλαίσια της συζήτηση για τη Ρουμανία στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σαν ε, τι θα γίνει με αυτόν τον πίνακα και πώς θα ε, τον χρησιμοποιήσετε. Το άλλο θέμα που θέτω αφορά τους Ρωμά. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί τον τελευταίο καιρό και από την Διεθνή Τράπεζα και από ε, άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ε, δεν έχουν όμως τύχη της απαιτούμενης, ε, θα έλεγα, δημοσιότητας Καλό θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας όπως της Παγκόσμιας Τράπεζας, συγγνώμη, όπως επίσης και τα στοιχεία της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη του UNDP. Πώς ερμηνεύετε τα δεδομένα αυτά και πώς χρησιμοποιείτε τα δεδομένα αυτά στον διάλογο τον οποίο έχετε με τα κράτη-μέλη και πώς μπορείτε εσείς να προβλέψετε τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής για τους Ρωμά. Κυρία Ιντβέλτ, Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ρέντινγκ, όπως και ο κύριος Δρούτσας το έκανε, το λεπτομέρειες για το πακέτο αυτό για τα δεδομένα. Έχει δύο σκέλη, αλλά μόνο το ένα κινείται φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο τώρα έχει ξεκινήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται η ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτά σκέλη έχει κλονιστεί. Για μένα θα ήταν αδύνατο να υιοθετήσω οποιοδήποτε μέτρο για την αστυνομική συνεργασία αν δεν συνοδεύεται από σωστούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Πώς το βλέπει η Επίτροπος αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα επιπλέον στοιχεία για τη διεθνή διάσταση της προστασίας των δεδομένων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί στην παρούσα φάση. Ήδη σε αυτή τη φάση ε, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και ε, θα έλεγα ε, χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες και όχι μόνο τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και μεγάλες άλλες χώρες εταίρους εμπορικές, εμπορικούς συγγνώμη όπως η Κίνα, η Ινδία κτλ. Τώρα για το πιο πρόσφατα το θέμα της απέλασης των Ρωμά από τη Γαλλία. Θα ήθελα να μάθω αν η Επίτροπο σκοπεύει να κάνει κάποιες προτάσεις και να μας πει επίσης ε, τι θα κάνει και με ε, τον οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και όλων των συναφών κατηγοριών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, βεβαίως με τη Γαλλία, τι συμβαίνει εκεί πέρα και τι θα κάνουν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά. Μετά, και πάλι για τους Ρωμά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε τι ακριβώς θα γίνει με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα προγράμματα συνεργασίας. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, όπως ε, η τροποποίηση των επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων, καλύτερες ε, και πολυδιάστατες προσεγγίσεις. Θα συμπεριληφθούν όλα αυτά στην έκταση πρόοδους και πότε θα γίνει αυτό για τους Ρωμά και μετά ο ρόλος των Task Force. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι η Γενική Διεύθυνσή σας παραβλέπει ε, επιβλέπει ε, την ε, ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά. Αναδεικνύονται στοιχεία τα οποία γενικώ δεν είναι γνωστά. Εκεί η Task Force μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και σήμερα το πρωί στην έκθεση της κυρίας Δάνοκα... Ε, για τον ε, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, κύριος οργανισμός προάσπισης των δικαιωμάτων των Ρωμά. εξετάσαμε λοιπόν αυτή την έκθεση σήμερα και είπαμε ότι τα καθήκοντα του οργανισμού αυτού ήδη υπερβαίνουν τις δυνατότητές του. Αυτό συμβαίνει και με το ζήτημα των Ρωμά. Ήδη από πέρσι φάνηκε πόσο σημαντική είναι η καλύτερη ε, παρακολούθηση. Ε, πολλά μπορώ να σας πω και για τη Γαλλία. Γι' αυτό θα ήταν καλό να το εξετάσετε. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πρώτο σχόλιο δεν πρέπει να το καταλογίσετε στο χρόνο που μου δίνετε γιατί εγώ ήθελα να ζητήσω το λόγο και στον πρώτο γύρο και σας ζήτησα χρόνο και όταν ο πρώτος γύρος καταλα... καταλαβαίνει μια ώρα και ένα τέταρτο και ο δεύτερος μονάχα το υπόλοιπο δεν μπορώ να επανέλθω στο θέμα αυτό αλλά χρησιμοποιώντας αυτά που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη... θα ήθελα να μιλήσω για τις διασφαλίσεις σε δικονομικό επίπεδο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απάντηση που δεν δώσατε κυρία Ρέντινγκ για το αν πραγματικά η απόφαση για τα θέματα αυτά θα ληφθεί μέσα σε αυτήν την θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για την νομική αρρωγή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το πακέτο των ε, <clears throat> δικονομικών εγγύσεων ήταν ένα πακέτο και ο στόχος του ήταν να υπάρχει μια ενιαία οδηγία σε σχέση με όλες αυτές τις διασφαλίσεις. Τώρα Έχουμε διασπάσει αυτό σε μια οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο και σε μια οδηγία για την νομική αρρωγή. Κατανοώ, όπως λέτε, ότι είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Αλλά η Κομισιόν έχει στα χέρια της μελέτες που αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα του θέματος αυτού, αυτό που θα θέλαμε ήταν να μπορέσει να υπάρχει μια ενιαία εφαρμογή του δικαίωματος που, που απορρέει από την Χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων να υπάρχει και νομική αρρωγή και πρόσβαση σε δικηγόρο. Αν εμείς έχουμε μονάχα την πρόσβαση σε δικηγόρο χωρίς νομική αρρωγή, αυτό σημαίνει ότι πολλοί πολίτες δεν θα μπορούν να υποφεληθούν αυτού του δικαιώματος. Επίσης αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για, για το ευρωπαϊκό ένταλμα ε, σύλληψης είναι ανισχυτικό. Γιατί τότε τι αποφάσει θα πάρει η Κομισιόν ω θεματοφύλακα των συνδικών μετά από αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, τι θέση θα πάρει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν προβλέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί ακριβώ αυτό το πρόβλημα με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Ήθελα να σα πω και κάτι άλλο, ίσω δεν έχω χρόνο, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε εσά για το θέμα τη βία κατά των γυναικών. το, πρόγραμμα προπολογισμού για τα δικαστικά θέματα, όπω είπατε στην παρέμβασή σα στην Ολομέλεια, δεν υπάρχει ένα χωριστό τμήμα που έχει να κάνει με την προστασία των θυμάτων. Υπάρχει το πρόγραμμα Δάφνη, αλλά κυρία Ρέντινγκ, πρέπει να σα πω ότι ενώ χαιρόμαστε για την παρουσίαση για το πρόγραμμα υποστήριξη των θυμάτων, το πρόγραμμα Δάφνη έχει τα ίδια χρήματα που είχε στο προηγούμενο πολίτε πλαίσιο. Δεν έχει αυξηθεί δηλαδή το ποσό το οποίο δίδεται στο πρόγραμμα Δάφνη από το έτος 2007. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη μνήμα για την πρόληψη της τοξικονομίας, τοξικομανίας συγγνώμη, που είναι θέμα δημόσιας υγείας, αλλά ίσως θα έπρεπε να δώσετε την ίδια και περισσότερη έμφαση στο θέμα της βίας κατά των γυναικών από ότι το οποίο προβλέπεται ήδη να αντιμετωπιστεί στο στο πακέτο κατά των θυμάτων, υπέρ των θυμάτων, αλλά δεν τη χάνει χρηματοδότηση. Κυρία Ρομέρο, η Προεδρία της Επιτροπής είναι που αποφασίζει την κατανομή του χρόνου. Όταν η Κομισιόν έχει να παρουσιάσει ένα μονάχα θέμα, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να εξασφαλίσουμε μια ε, ένα γύρο μονάχα ερωτήσεων και απαντήσεων και να καλύψουμε όλα τα θέματα όταν υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση τρία τουλάχιστον διαφοροποιημένα θέματα στην παρέμβαση κυρία κυρίας Επιτρόπου νομίζω ότι έχει κάθε νόημα να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τη συζήτηση για να μην αναμειγνύονται τα διάφορα σημεία και να μπορεί να απαντήσει η κυρία Επίτροπος με έναν τρόπο ο οποίος να είναι σαφής. Δεν μπορεί να υπάρξει μια απάντηση συλλήβνη σε όλα τα θέματα. Ναι, πράγματι λέτε ότι κράτησε ένα χρόνο και τέταρτο ο πρώτος γύρος και τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν θέματα, τα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των Ρωμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τάθηξε η κυρία Επίτροπος. Αλλά δεν νομίζω ότι ε, έχει την δυνατότητα, έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται κάποιος ότι δεν τον άφησα να, του, να λάβει το λόγο γιατί δεν του έδωσε το λόγο. Εγώ πάντα προσπαθώ με τη μεγαλύτερη ευκαμψία να εξασφαλίσω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους. Επιμένω πάντα στην ανάγκη να τηρήσουμε ένα χρόνο σε κάποιο βαθμό που συναρμόζεται με την μέση διάταξη και να σεβαστούμε και το χρόνο των άλλων. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Επιτροπή μα και στην Ολομέλεια ένα βουλευτή ο οποίο θέτει το ερώτημά του μετά λέει ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος πριν λάβει το λόγο και μόλις λάβει το λόγο δεν περιμένει την απάντησή του και φεύγει. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία. Δίνω το λόγο στην κυρία Μορβάη μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πέμπτη ή έκτη φορά που συνοψίζω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι η, το μεγαλύτερο σοκ για μένα στην ανθρώπινη ιστορία σε ό,τι αφορά την ε, αστυνομική συνεργασία ε, για τα δικαστικά ζητήματα και χαίρομαι που συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου. Ζητώ συγγνώμη που ε, από τους συναδέλφους που έχουν ξανακούσει αυτή την ιστορία αναφέρομαι σε μια ε, υπόθεση Ιρλανδής υπηκόου που ήρθε στην Ουγγαρία και, και χτύπησε με το αυτοκίνητό της δύο παιδιά, δύο και πέντε ετών που περίμεναν με τη γιαγιά τους ε, στο πεζοδρόμιο και, και η οικογένεια έχασε έτσι δύο παιδιά λόγω της ε, απίστευτα πρόσεχτης οδήγησής της και τα δύο παιδιά λοιπόν έχασαν τη ζωή τους. Ε, η Ουγγαρία επέτρεψε στην Ιρλανδία Πίκο να επιστρέψει στη χώρα της, ε, για να το πω απλά με εγγύηση και την καταδικάσαμε σε τριετή κάθριξη. Αυτό το άτομο τώρα βρίσκεται στην Ιρλανδία και δεν ε, ούτε έχει απελαθεί ούτε εκτελείται η ποινή. Επομένω αυτό το πρόσωπο κυκλοφορεί ελεύθερο και δεν έχει τιμωρηθεί το έγκλημα. Εσείς, Επίτροπε, με το Ουγγρικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, πέρσι και μάλιστα όλες οι εφημερίδες ήταν ε, γεμάτες ε, με φωτογραφίες σας. Τι πετύχατε λοιπόν εκεί πέρα και εσείς ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των θυμάτων τι έχετε να μας πείτε και τι έχετε να πείτε στους γονείς. Έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο για να κινήσουν μια διαδικασία. Επαναλαμβάνω το ερώτημα της ε, κυρία Γκάλ. Μπορούν να προσφύγουν στο δικαίωμα του Λουξεμβούργου ή του Στρασβούργου και εσείς ως ε, επικεφαλής και ε, προεξάρχουσα προσωπικότητα σε αυτόν τον τομέα. Τι έχετε να μας πείτε και τι έχετε να κάνετε. Έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο στο ευρωπαϊκό σύστημα εσείς που θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντικό να ε, εκπροσωπούνται τα, τα, και να προσπιζόμαστε τα δικαιώματα των ε, θυμάτων. Η κυρία Ζίπελ. Κατανοώ ότι υπήρξε πρόβλημα με το χρόνο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Ακόμα και τέσσερις ώρες να είχαμε, δεν θα φτάνε πάλι ο χρόνος. Εμείς, σαν ε, βουλευτές, θα πρέπει να έχουμε κάποιον αυτοπεριορισμό και να περιοριζόμαστε στα θέματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, αλλιώ δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε, να έχουμε μια απάντηση όλοι στην στο ερώτημά μα. Εγώ νομίζω ότι σε όλη τη συζήτηση υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρω. Τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ωραία, το είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, όταν μιλάμε για τι διαδικασίε και τι διασφαλίσει. Εμεί συζητήσαμε <clears throat> στο θέμα τη Ευρωπόλ ότι εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε επεξεργασίε στοιχείων και στον τομέα τη δικαιοσύνη αλλά όταν πρόκειται για τα θέματα προστασίας των δεδομένων, τα κράτη-μέλη μας τροχοπεδούν πάντα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αυξήσουμε τη πίεση στα κράτη-μέλη. Τι κάνει η Κομισιόν να μας πει γιατί δεν προχωράμε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων των ε, υπόπτων ή κατηγορούμενων. Δεν μπορούμε συνέχεια να δημιουργούμε περισσότερες ε, δυνατότητες συλλογής δεδομένων, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, και μετά να αγνοούμε τα, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων ή των θυμάτων. Πρέπει η Ευρώπη, να το καταλάβουμε αυτό, η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει μονάχα όταν τα κράτη-μέλη βοηθούν την Ευρώπη και όχι όταν την τροχοπέδουν. Στην ε, απάντηση τώρα στο... στην κυρία Πίτροπο έρχομαι για να απαντήσει. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε. Όπως κάνω συνήθως και ελπίζω να το αναγνωρίσετε, προσπαθώ να απαντήσω με σοβαρό τρόπο και δεν χρησιμοποιώ ξύλινη γλώσσα. Για την προστασία των δεδομένων λοιπόν. Εδώ το σχέδιό μου είναι σαφές. Θα δώσω μάχη για το πακέτο Βεβαίως, ορισμένα κράτη-μέλη διστάζουν με την πρότασή μας. Βεβαίως και ορισμένες χώρες προσπάθησαν από την αρχή να ξεχωρίσουν την οδηγία και να μείνει μόνο ο κανονισμός προς εξέταση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σταματήσαμε στην επίσημη συνάντηση, στην ανεπίσημη συνάντηση, συγγνώμη, όπου ήταν παρόν και ο πρόεδρός σας, το ανεπίσημο συμβούλιο εννοεί η Επίτροπος. Και για μας και για σας ήταν ανέκαθεν σαφές ότι μιλάμε για δύο αντίστοιχα επίπεδα δικαιωμάτων και σε επίπεδο ιδιωτικό και σε επίπεδο εμπορικό και σε επίπεδο δημόσιο-κρατικό. Η συνθήκη δεν κάνει καμία διαφοροποίηση. Συνεπώς εμείς εφαρμόζουμε την συνθήκη απλά και δεύτερον θα πρέπει να διευρύνουμε την ισχύ της οδηγίας και στην εσωτερική εθνική ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων άμεσα σε διαφορετικές αρχές. Αυτό ορισμένες κυβερνήσεις ε, του ε, το ασκούν πολύ σοβαρή κριτική. Όταν βέβαια συζητάω με εκπροσώπους του νόμου από τις διάφορες χώρες μου λέγουν ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δεδομένα τα οποία είναι καθημερινά και τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμεθοριακή θα έλεγα χρήση. Θα ήταν λοιπόν παράλογο να προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε ένα διαχωρισμό και οι δύο μορφές των δεδομένων πρέπει να υπακούν στους ίδιους κανόνες και δεν κατανοώ τις απόψεις ορισμένων υπουργών εσωτερικών που θέλουν να επιβαρύνουν διοικητικά τις αρμόδιες αρχές τους χωρίς να σέβονται τη συνθήκη. Λοιπόν, διευκρίνησα και εγώ, διευκρινήσατε και εσείς νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να συνεχίσουν έτσι με συνδυασμένο τρόπο. Τώρα έρχομαι στο θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εάν πράγματι υπάρχει ένα θέμα όπου το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με το Συμβούλιο είναι αυτό. Όταν συντάσσει κανείς μια νομοθετική πράξη, θέλει να συντάξει την βέλτιστη δυνατή και άμεσα εφαρμόσιμη. Όταν συντάσσει κανείς έναν κανονισμό, ο οποίος είναι άμεσα εφαρμόσιμος, και ξέρετε ότι δυσκολία θα έχουμε εμείς ε, έτσι ώστε η πρότασή μας να είναι άμεσα εφαρμόσιμη, δεν θέλει να επανέρχεται στο συγκεκριμένο θέμα αναεξάμεινο και να μεταρρυθμίζει τις νομοθετικές επιμέρους ρυθμίσεις. Θα πρέπει δηλαδή η πρότασή μας να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς κάθε φορά να, να χρειάζεται ε, μία πλήρης μεταρρύθμιση. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα ακριβώς τις εφαρμοστικές διατάξεις και τις αρμοδιότητες τις εφαρμοστικές και τις οι πράξεις που περιλαμβάνουν στις, περιλαμβάνονται στη συνθήκη. Δεν τις φανταστήκαμε εμείς για να αυξήσουμε τις δικές μας εξουσίες. Αν δείτε πού εμείς έχουμε εντάξει τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, θα διαπιστώσετε ότι κάθε φορά που το κάνουμε δεν το κάνουμε για σημαντικά θέματα ή για στρατηγικά θέματα. Αυτά αντιμετωπίζονται με συνολικότερο τρόπο. Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το τι είναι κάποια στρατηγικά θέματα, στρατηγικά στοιχεία, γιατί κάτι που εγώ θεωρώ στρατηγική σημασίας, εσείς μπορείτε να διαφωνείτε. Πάντως στις προτάσεις που κάνουμε ξεκαθαρίσαμε ότι σημαντικά θέματα ή ε, στρατηγικά θέματα δεν καλύπτονται από τις νομοθετικές αυτές κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά τεχνικά θέματα τα οποία απαιτούν άμεση απόκριση. Κοιτάξτε τι λέει η καινούργια συνθήκη. Οι κατεξουσιοδότηση αυτές πράξεις μπορεί να αποφασιστούν μόνο επί τη βάση της συνθήκης, σεβόμενη τη νομική ρύθμιση και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Όχι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια γωνία μόνη της θα μαστιγώνει τους ε, πολίτες. Όχι, αυτό γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα κουτί. Ας το συζητήσουμε το πλαίσιο αυτό και θα μου πείτε αν έχουμε προχωρήσει υπερβολικά ή αν πράγματι αυτό το οποίο προτείνουμε έχει νόημα. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Προσπαθήσαμε να μην περάσουμε λοιπόν την κόκκινη γραμμή. Ε, κάθε τι το οποίο θεωρείται σημαντικό και ουσιώδες ε, περιλαμβάνεται στον κανονισμό και δεν υφίσταται την διαδικασία <clears throat> των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Γνωρίζω αυτό το οποίο είπατε για τις τρίτες χώρες και ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να έχουμε ισχυρούς ευρωπαϊκούς νόμους είναι για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με τα υπόλοιπα τμήματα του κόσμου σαν μια ήπειρος με υπηρετικούς κανόνες. Γιατί αν το κάνουμε αυτό στα γαλλικά ονόρο δισπερσέ, με πολυδιάσπαση δηλαδή, τότε το αποτέλεσμα σίγουρα δεν θα είναι θετικό. Αυτό είναι ακριβώς το λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε αυτού του είδους τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα, τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά όργανα, τι θα γίνει με το Eurojust κτλ. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη σε αυτό. Πρώτον, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από κανονισμούς. Αυτή αυτή στιγμή έχουμε τη νομική ε, ρύθμιση στη διάθεσή μας, θα προσαρμόσουμε τους κανονισμούς. Αυτό είναι σαφές. Και το ίδιο ισχύει επίσης και για υπηρεσίες όπως η Europol. Ήδη στην ανακοίνωσή μας ε, στις αρχές του 12 είπαμε ότι θα ξεκαθαρίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους πριν το τέλος του χρόνου δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις δηλαδή στους γενικά εφαρμόσιμους κανόνες για όσους εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους όσους θέλουν να είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για το ένταλμα σύλληψης. γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεων, κοινοτικό επίπεδο αποφάσεων και να μην αρκεστούμε σε διακυβερνητικές, σε διακυβερνητικές αυστηρά αποφάσεις. Αυτό το θέλουμε ακριβώς για να μην υπάρξει διαφορετική ερμηνεία και διαφορετική εφαρμογή του νόμου. Κάτι τέτοιο θέλουμε να το αποτρέψουμε. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό. Είμαι ανυπόμονη βέβαια, αλλά μόνο εδώ και δύο χρόνια μπορέσαμε να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ό,τι είχε αποφασιστεί στο παρελθόν ήταν αμυγός διακυβερνητικό και οι περισσότερες από τις κριτικές που μας απευθύνονται εδώ είναι κριτικές που θα πρέπει να στραφούν στα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη βασίζονται ακριβώς στις διακυβερνητικές συμφωνίες και αυτές οι συμφωνίες όπως βλέπουμε λειτουργούν με ατελέστατους τρόπους. Είναι πως λοιπόν το καλύτερο που μπορώ εγώ να κάνω στην περίπτωση αυτή είναι να λειτουργήσω σαν ενδιάμεσος ανάμεσα σε δύο αντιτιθέμενες απόψεις δύο διαφορετικών κρατών μελών. Και δεν μπορώ να πιέσω τις χώρες αυτές να προχωρήσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Για να το πετύχω αυτό απαιτείται ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθεσίας. Και γι' αυτό ακριβώς θέτουμε τα πάντα τώρα στα πλαίσια ευρωπαϊκής νομοθετικής τάξης. Και γι' αυτό ακριβώς και από το 2014 θα προχωρήσουμε στην λεγόμενη σε εισαγωγικά λισαβονοποίηση όλων αυτών των διακυβερνητικών κανόνων. Έχουμε πολλές φιλοδοξίες προς την κατεύθυνση αυτή, τώρα θα δούμε πώς θα το πετύχουμε, γιατί όταν το πετύχουμε αυτό σημαίνει ότι αυτόματα όλες οι διακυβερνητικές συμφωνίες θα μετατραπούν σε συμφωνίες ή σε δίκαιο μάλλον ευρωπαϊκό. Θα υπάρξουν πάρα πολλές συζητήσεις από ό,τι φαίνεται με τα κράτη-μέλη σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα για τα κριτήρια της Κοπενχάγης. το θέμα της λειτουργίας του δικαστικού σώματος, το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων, το θέμα της καταπολέμησης της διαφοράς, όλα αυτά είναι θέματα που είναι σε κρεμότητα. Όπως είπα Όταν οι χώρες αυτές ε, γίνουν κράτη-μέλη, γίνουν μέλη, ε, τότε θα μπορέσουμε να δράσουμε. Και τότε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Και γι' αυτό ακριβώς πρότεινα μια σταδιακή, θα έλεγα, εφαρμογή αυτού του πίνακα επιδόσεων. Ο λόγος ε, είναι ακριβώς ότι η εμπιστοσύνη στο σύστημα το δικαστικό θα βοηθήσει και στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εντάξουμε αυτό το scoreboard, τον πίνακα επιδόσεων, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτή τη στιγμή συγγίνει αυτό, τότε σε μια δεύτερη φάση θα μπορέσουμε το σύστημα αυτό να το αναπτύξουμε και σε δικαστικό επίπεδο και για τα υπόλοιπα στοιχεία της λειτουργίας της δικαιοσύνης, τα οποία δεν συνδέονται αποκλειστικά με την οικονομική δραστηριότητα. για το τα ζητήματα Σέγγεν. Έχει φύγει ο συνάδελφος, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα πω. Γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και είναι σημαντικό το θέμα. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή κάνει τεχνική ανάλυση για να δει εάν ένα κράτος μέλος έχει προετοιμάσει τεχνικά τα σύνορά του για να ενταχθεί στο σύστημα Σέγγεν. Ουσιαστικά δηλαδή περισσότερο αν τα εξωτερικά σύνορα είναι από τεχνική πλευρά ε, καλά προστατευμένα. Αυτό το έργο έχει γίνει και η Επιτροπή έχει πει ξεκάθαρα ότι τα δύο εν λόγω ε, κράτη-μέλη, Βουλγαρία και Ρουμανία, είναι μια χαρά από τεχνικής άποψης. Η πολιτική απόφαση λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη. Με ομόφωνη απόφαση. Και όχι για τις τεχνικές πλευρές, αλλά από την πολιτική σκοπιά. Και εκεί φαντάζεστε και το βλέπετε. Το είδατε στην υπουργική διάσκεψη ότι έχει ακυρωθεί, Φαντάζεστε λοιπόν τι είδους ε, πολιτική συζήτηση ε, διεξάγεται αυτή τη στιγμή ε, για την συνέχιση της ε, Σέγγεν. Θα θίξω το θέμα των Ρωμά τελευταίο. Για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο οργανισμός στη Βιέννη και επιτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο που με βοηθάει και εμένα προσωπικά γιατί δεν γνωρίζω όλες αυτές τις πληροφορίες και λεπτομέρειες. Χρειάζομαι λοιπόν αυτές τις ε, τεκμηριωμένες ε, αναλύσεις και τα δεδομένα που λαμβάνουμε από αυτόν τον οργανισμό. υπάρχει διαφωνία με κάποια κράτη-μέλη για τον τρόπο λειτουργίας ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ε, του προγράμματος εργασιών του. Ξέρετε ότι κάτι μέλη πρέπει στο Συμβούλιο να υιοθετήσουν ομόφωνα το πρόγραμμα ε, εργασίας του οργανισμού πρόσφατα. Έχουν αρνηθεί να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα εργασίας του ΦΡΑ ε, θεματικού τομεί όπω η αστυνομική συνεργασία, δικαστική ε, συνεργασία σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο. Και εγώ έχω το δικαίωμα ε, να ζητήσω από τον οργανισμό αυτό να επιτελέσει αυτά το καθήκοντα. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε κάποιες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα Δάφνη. Πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να σταματήσει το πρόγραμμα αυτό. Προτείνει να συνεχιστεί ε, στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιωμάτων και ηθαγένειας. Έχουμε το πρόγραμμα Δάφνη, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, ηθαγένειας και ε, του θεματολογίου ισότητας και κατά των διακρίσεων. Με στόχο να έχουμε συνέργειες για την απλούστευση της διαδικασίας, για να έχουμε περισσότερους πόρους ε, στη συνέχεια. Να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα από τα λίγα προγράμματα που ε, βγαίνουν από την Επιτροπή χωρίς μείωση. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Άλλο θέμα αυτό. Άρα όμως η Επιτροπή για όλα αυτά τα προγράμματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, την ηθαγένεια, τις γυναίκες και ούτω καθεξής, δεν έχει υπάρξει μείωση. Και για να σας θέσω ακόμα έναν ειδικό στόχο στο Δάφνη για το πρόγραμμα δικαιωμάτων και θαγένειας αν θέλετε μάλλον να συμπεριληφθεί ακόμα σε ένας ειδικό στόχος, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν θέλαμε αρχικά να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι και αιτία πολέμου. Αν το επιθυμούν αυτό οι συνομοθέτες, θα το κάνουν. για τους ομοφυλόφιλους λεσβείες, τα μεθυλιακά άτομα και ούτω καθεξής ε, και για τον αντίστοιχο οδικό χάρτη. Ξέρετε ότι ε, η αρχή των μη διακρίσεων ε, λόγω φύλου και σεξουαλικών προτιμήσεων είναι βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Έχουμε κινήσει διαδικασίες παραβάση εναντίον κάποιων κρατών μελών που δεν έχουν υλοποιήσει σωστά την οδηγία ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Και αυτό έγινε και όταν υπήρχε τέτοια διάκριση. Και δεύτερον, συγκεκριμένη πρόταση στον ε, τομέα ε, αστικού δικαίου, να δοθεί το δικαίωμα σε όλα τα ζευγάρια. Αν δείτε, οι προτάσεις μου είναι ουδέτερε ως προ τη διάσταση του φύλου. Δίνεται λοιπόν το δικαίωμα σε όλα τα ζευγάρια. Ε, τα ζευγάρια. Για παράδειγμα, το γαμικό ιδιοκτησιακό καθεστώ, για παράδειγμα. Αυτή είναι η αρχική πρόταση. Μετά πρέπει να γίνει συζήτηση Κοινοβουλίου-Συμβουλίου. Για το ζήτημα της ε, νομικής αρρωγής. Έχω ήδη εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε και γιατί χρειαζόμαστε αυτή την ανάλυση. τις μελέτες. Να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ακόμα μελέτη και βάσει των όσων έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να καταθέσουμε νομική πρόταση. Θέλω όμως να το κάνω αυτό, την έχω γράψει, έχω δεσμευτεί ότι θα το κάνω το 2013. Περνάω στους Ρωμά. Ναι. Η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πλήρως ή ικανοποιητικά εφαρμόσει <clears throat> τις εθνικές στρατηγικές για τους Ρωμά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα ενσωμάτωσης αυτού του πληθυσμού, το οποίο είναι μακριά από το να έχει επιληθεί. Και τα παιδιά των Ρωμά δεν έχουν ακόμα παρουσία στα σχολεία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει, από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να δεν θέλουμε το πρόβλημα να διαιωνιστεί και να ακολουθεί τις επόμενες γενιές το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, είχα πολύ σοβαρές συζητήσεις με τον ε, ομολόγο συνάδελφό μου στη Γαλλική Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εσωτερικών, επί τη βάση των συνομιλίων αυτών. Ο νέος γαλλικός νόμος για την ελεύθερη κυκλοφορία τελικά εφαρμόστηκε. Αυτό δεν επιλύει από μόνο του το πρόβλημα της ενσωμάτωσης στο Ρωμά. Αυτό αφορά μονάχα τα <clears throat> μεμονωμένα δικαιώματα ενός Ευρωπαίου πολίτη να μην απελάβνεται από ένα κράτος μέλος χωρίς δικαστική απόφαση και χωρίς την δυνατότητα να αντιταχθεί σε ένα τέτοιο μέτρο και να γίνει ακουστή η άποψή του και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό σαν μεμονωμένη περίπτωση ενώπιον των δικαστηρίων. Γι' αυτό θα γίνουν ορισμένες ενέργειες πρώτα απ' όλα. Η ανάλυση και επεξεργασία των εθνικών στρατηγικών Ρωμά θα λάβει χώρα, όπως έχω υποσχεθεί. Θυμάστε ότι την τελευταία φορά σας είχα παρουσιάσει τη στρατηγική που έχει προτείνει κάθε κράτος μέλος για την αντιμετώπιση των Ρωμά και είπαμε θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση του τι γίνεται σε κράτος μέλος. Αυτή η ανάλυση γίνεται ανά κράτος μέλος, θα περατωθεί αυτή η διαδικασία. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτό δεν επαρκεί και γι' αυτό το λόγο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν έλαβαν χώρα και όλα αυτά τα γεγονότα και πάλι, με διαφορετικό τρόπο αλλά Παρ' όλα αυτά συνέβησαν. Πρότεινα μία προσέγγιση που συνίσταται σε τρία βήματα. Πρώτα απ' όλα, τον Οκτώβριο τα εθνικά σημεία επαφής με, για τους Ρωμά θα συναντηθούν. Ξέρετε ότι είχαμε καθορίσει ένα εθνικό σημείο επαφής για τους Ρωμά μετά από την πρώτη κρίση θα συναντηθούν εδώ στις Βρυξέλλες για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχει επιτευχθεί πρόοδος, αν δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, πού δεν λειτουργούν τα πράγματα καθόλου και ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, κατά πόσο τα κονδύλια απορροφώνται ή όχι, ποιες είναι οι υποσχέσεις που έχουν γίνει στο χαρτί και τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δεύτερο στοιχείο, όταν έχουμε συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα πρωτοπόρων κρατών μελών. Με τρία ειδικά των μελών σε αυτή την ομάδα πιονιέρων κατά κάποιο τρόπο χώρες που έχουν μεγάλο πληθυσμό Ρωμά στο έδαφος τους. Δεύτερον, κρατάει μέλη που έχουν κάνει ενδιαφέρουσες δράσεις ενσωμάτωσης των Ρωμά, όπως η Φιλανδία, παραδείγματος χάρη. Όχι αυτές που θα σκεφτόσασταν. Και τρίτον, τα κράτη-μέλη που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Να έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες λοιπόν χωρών να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βοηθήσουμε το εθνικό επίπεδο για να προχωρήσει περαιτέρω. Και τρίτο βήμα, επί τη βάση της εργασίας αυτής, εάν υπάρχει ανάγκη, είμαι έτοιμη να κάνω και κάποια σύσταση. Σας ευχαριστώ, λέει Νομίζω ότι κάνετε μια προσπάθεια να καλύψετε εγκαίρως όλες τις ερωτήσεις. Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα την προσπάθειά σας να είστε συνοπτικοί και να καλύψετε όλα τα ερωτήματα τα οποία σας ετέθησαν. Είναι προφανές ότι όταν η Επίτροπος Ρέντιν παρίσταται στην Επιτροπή Λίμπε τότε θα προκύψει μια συζήτηση. Θα υπάρξει μια ευρύτατη συζήτηση. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να έρχεστε πιο συχνά εδώ. Και έτσι θα υπάρχει κατάλληλη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση για την Ουγγαρία.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 So, so let's go. Let's go. Well, now, final point, 45 minutes. Τελευταίο σημείο 45 λεπτά. 6 παρατέταρτο κανονικά πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση αυτή για τα μέτρα και τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ουγγαρία. Πρόταση που κατετέθη το Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλούμεθα λοιπόν τώρα να ακούσουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα μας δώσει ο εισηγητής. Έχει ήδη συνταχθεί το κείμενο εργασίας από τον κύριο Ταβάρες. Και όλοι γνωρίζετε ότι θα υπάρξει και μια επίσημη αντιπροσωπεία, μια αντιπροσωπεία ad hoc που είναι κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο θα επισκεφθεί την Ουγγαρία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Αντιπροσωπεία λοιπόν στην Ουγγαρία ad hoc. Αυτό δεν είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τους κανόνες των τακτικών αντιπροσωπιών που στέλνουμε τακτικά στο εξωτερικό από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι κάτι διαφορετικό, πρόκειται για μια αντιπροσωπεία ad hoc επτά συν ένας, πρόεδρος ο ένας. Θα επισκεφθούμε τη Βουδαπέστη. Θα έχουμε επαφή με συνομιλητές, εκπροσώπους θεσμικών οργάνων, εκπροσώπους ΜΚΟ της κοινωνίας των πολιτών και θα μπορέσουμε έτσι να δούμε πώς είναι τα πράγματα επιτόπου και θα γυρίσουμε στις Βρυξέλλες για να διατυπώσουμε την τελική μορφή της έκθεσης την οποία αναλάβαμε σαν υποχρέωση να φέρουμε εις πέρα τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Δεν συζητάμε λοιπόν σήμερα για να εξαντλήσουμε το θέμα, για να εμβαθύνουμε μεμονωμένα, αλλά για να δούμε ακριβώς πώς έχει προχωρήσει στην προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όχι από την στιγμή που ξεκινάει η συζήτηση για την Ουγγαρία, αλλά από την αρχή τη συζήτηση για αυτή την έκθεση είχαμε πει, είχαμε υποσχεθεί να συζητήσουμε πρώτα και να συμφωνήσουμε για τη μεθοδολογία και μετά να περάσουμε στο περιεχόμενο. Μεταξύ τη μεθοδολογία και του περιεχομένου, βέβαια, υπάρχει η εξέβρεση των συγκεκριμένων στοιχείων. Αυτό θα γίνει στη Βουδαπέστη από την αποστολή μα την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό τμήμα της έρευνας των πραγματικών στοιχείων που πρέπει να γίνει στα πλαίσια αυτής της έκθεσης ώστε να καταλήξουμε σε έγγραφα εργασίας. Τα έγγραφα αυτά εργασίας ανταποκρίνονται σε μία άλλη υποχρέωση που έχουμε αναλάβει ότι πρέπει να είναι εξισορροπημένα και να περιλαμβάνουν και τις συμβολές όλων των πολιτικών ομάδων, φυσικά να βασίζονται στα πραγματικά γεγονότα, αλλά να λαμβάνουν υπόψη και τις θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων. Με ένα ανοιχτό και διάφορο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά εργασία, τουλάχιστον τα δύο τα οποία έχουν συνταχθεί μέχρι τώρα, θα πρέπει επίσης να λειτουργήσουν και ως προπαρασκευαστικά έγγραφα για την αντιπροσωπεία μας προς τη Βουδαπέστη, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν με τις περισσότερο πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από την αποστολή μας. Το πρώτο έγγραφο το έχω συντάξει μαζί με τον Φρανκ Έγγελ από κοινού και αφορά το δικαστικό σύστημα στην Ουγγαρία και το δεύτερο έγγραφο που έχουμε τώρα ενώπιόν μας είναι το έγγραφο για τα θεμελιώδη δικαίωματα και τις θεμελιώδεις αξίες που έχει γίνει από τον πρόεδρό μας και τον σκιώδη εισηγητή για το θέμα αυτό. Τα επερχόμενα έγγραφα εργασία θα συζητηθούν με τον εισηγητή και είμαι ανοιχτό να ακούσω προτάσει και να δεχτώ τι προτάσει για τα έγγραφα εργασία. Υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, το οποίο και αυτό θα συνταχθεί μαζί με τη Ρενάτε Βέμπερ καθώς προχωρούμε για αυτήν την ε, έκθεση και επίσης και άλλα ε, έγγραφα εργασίας μπορούν να συνταχθούν ακόμα και μετά από την επίσκεψή μας. Πρέπει μάλιστα να συγγραφούν μετά την επίσκεψή μας στην Ουγγαρία. Είναι απεξηραμένα έγγραφα αυτά, δεν έχουν σχόλια ή συμπεράσματα και αυτό είναι θεληματικό βασίζονται σε νομικά κείμενα που είναι τα θεμελιά της εργασίας μας, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Συνθήκη και τα νομοθετήματα της Ουγγαρίας τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και τα οποία μας έχουν δοθεί από τις ε, Ουγγρικές Αρχές, ο Θεμελιώδης Νόμος και οι επιμέρους, οι επιμέρους νόμοι που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Βασιζόμαστε επίσης και σε στοιχεία που μας έχουν δοθεί από άλλους φορείς οι οποίοι επεξεργάζονται τα θέματα αυτά, όπως είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς έχουμε αντλήσει πολλά από τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και το πράττουμε και πάλι σε αυτό το έγγραφο. Επομένως έχουμε μια στέρεα βάση για το κείμενο το οποίο θέλουμε να εκπονήσουμε. Ξεκινούμε λοιπόν για, με το ερώτημα του ποιες είναι οι κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να έχουμε ασαφείς συνεφελώδες αξίες, βασιζόμαστε στις αξίες που αναφέρονται στις συνθήκες και αυτό το έγγραφο αναλύει κάποιους από τους ε, σημαντικούς νόμους και τις ε, πρόνοιες του Ουγγρικού Συντάγματος. Εκφράζει άποψη και κρίση για το αν έχουν να κάνουν παραδείγματος με θέματα αμοιβέ εμπιστοσύνη. Και ένα από τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε που είναι το θέμα της, του διαχωρισμού των εξουσιών. Δεν αντλούμε συμπεράσματα για το θέμα αυτό. Απλώς λέμε σε αυτό το στάδιο ότι είναι ακρογωνίας λήθος της δημοκρατίας ο διαχωρισμός των εξουσιών και βλέπουμε που είναι αυτή τη στιγμή τα όρια σε, τα οποία πορεύουν από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και επίσης αυτά που προκύπτουν από το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα. και επομένως είναι πολύ χρήσιμο για μένα να ακούσω τις απόψεις και όχι να συνεχίσω να μιλώ. Και ίσως ο πρώτος ως ε, συνεισηγητής για το σημείο αυτό, σαν συγγραφέας και αυτός ε, μαζί μου για αυτού του έγγραφου και οι άλλοι σχεδόν συζητητές θα ήθελαν ίσως να μου πούνε κάτι περισσότερο για το πώς θέλουν να προχωρήσουμε με αυτά τα έγγραφα και εγώ φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να πάρω τις αντιδράσεις σας και εγγράφος και να τις ενσωματώσω στο τελικό έγγραφο ως απόψεις της ΑΕΒ πολιτικής ομάδας. Προς το παρόν δεν έχω τίποτα άλλο να πω και θέλω να ακούσω την άποψη των συναδέλφων. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες. Όχι μόνο δεν έχω αντίρρηση, αλλά στηρίζω το έγγραφο εργασία γιατί ακολουθεί τις αρχές μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τον διαχωρισμό των εξουσιών, τις νέες ε, διατάξεις ε, για τα δικαστήρια και την συγκεκριτική αρχή. και τους νέους ε, κομβικούς νόμους που έχουν υιοθετηθεί <laughs> στην Ουγγαρία. Βεβαίω και παρακολουθούμε τι γίνεται με τον οδικό χάρτη ε, για την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχουμε ενώπιό μας ολόκληρο αυτό το θέμα που μένει να αναπτυχθεί όταν ολοκληρωθεί η αποστολή στην ε, Βουδαπέστη και, και συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σίγουρα θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω συζήτηση. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να ακούσουμε τα μέλη. Κύριε Άγγελ. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τους δύο που μας δώσατε το δεύτερο έγγραφο εργασίας, το οποίο όπως και το πρώτο αναφέρεται σε κάποιους τομείς οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν κάποια προβλήματα σχετικά με την θεμελιώδη νομοθετική ρύθμιση στην Ουγγαρία. Δεν περιμένουμε απαντήσεις στα περισσότερα από αυτά τα θέματα τώρα, αλλά για να μπορέσει το έγγραφο αυτό να είναι αντικειμενικό, πλήρως αντικειμενικό, θα πρέπει να δει κανείς τα πιθανά προβλήματα πώς μπορεί να αντισταθμιστούν από πιθανά πλεονεκτήματα. Πρώτον, ο έλεγχος του συνταγματικού χάρτη χωρίς διαβούλευση. Υπήρξε βέβαια στην Ουγγαρία διαβούλευση αρκετή πριν γίνει η αλλαγή στο Σύνταγμα. Ελήφθησαν από πλευρά των συνταχτών μαζικές προτάσεις πριν να καταλήξουν σε μια τελική απόφαση που έγινε δεκτή από τη Βουλή. Αλλά και πέραν αυτού θα πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, ότι οι συνταγματικές αρχές σε οποιοδήποτε κράτος, δηλαδή το Κοινοβούλιο, λειτουργήσε. Αν το Κοινοβούλιο ήταν εναντίον της πρότασης αυτής, δεν θα υπήρχε αυτό το νέο σύνταγμα. Το ότι το Κοινοβούλιο υπεψήφισε το σύνταγμα αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και πριν υιοθετηθεί το, κοινο, το σύνταγμα αυτό, υπήρξε μια μαζική λαϊκή διαβούλευση επί των διατάξεων του. Δεύτερον, το θέμα των κομβικών ή κεντρικών νόμων. Εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και θα το συζητήσουμε αυτό και την επόμενη εβδομάδα. Σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους των νόμων αυτών. Εγώ δεν νομίζω ότι εδώ ε, το πρόβλημα είναι ότι παραπέμπει το Σύνταγμα σε πάρα πολλού νόμους και στο δικό μου Σύνταγμα και σε άλλα Συντάγματα οι αναφορές αυτές ε, παραπέμπονται, υπάρχουν οι ρήτρες αυτές, παραπέμπονται σε επιμέρους νόμους. Το Σύνταγμα είναι ένας συνταγματικός χάρτης βασικός για τα θεμελιώδη. Και εδώ να συμπληρώσω, Πρόεδρε, κάποια επιπλέον στοιχεία για το τι σαν παράδειγμα το συνταγματικό δικαστήριο καλείται ή έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει. Όταν εγώ μελετούσα στο Βέλγιο α, τις αλλαγές στο Σύνταγμα μετά από την ομοσπονδοποίηση το 73-74, το δικαστήριο διαιτησίας στο Βέλγιο που ήταν στο ίδιο επίπεδο με το ανώτατο συνταγματικό ζήτησε ε, την αναθεώρηση τριών άρθρων. Το πρώτο, ισότητα των πολιτών μπροστά στον νόμο. Δεύτερο, ελευθερία στο σύστημα εκπαίδευσης. Και το τρίτο δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα από πολλά θα έλεγα που δείχνει ότι οι δυνατότητες αναθεώρησης και μεταρρύθμισης και οι τρόποι αναθεώρησης και μεταρρύθμισης είναι θέμα το οποίο μπορεί να διαφέρει κατά πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Και αν οι Ούγγροι επέλεξαν το συγκεκριμένο σύστημα, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα και αμφισβητήσιμο. Και μία τελική παρατήρηση, Πρόεδρε. Μία, θα έλεγα, λίγο τρομερή πρόταση ο προπολογισμό και η απόλυτη κυριαρχία του Ουγγρικού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό. Εμείς, αυτό εδώ το σώμα, πριν από λίγο καιρό αποφασίσαμε ότι η εθνική κυριαρχία στα δημοσιονομικά δεν υπάρχει πια. Αυτή τη στιγμή υπάρξει μάλιστα το σύμφωνο, το δημοσιονομικό. Κανένα κοινοβούλιο δεν θα ελέγχει τους προπολογισμούς όπως το παρελθόν. Κάποτε στη Γερμανία, όταν δεν λειτουργούσαν στα πλαίσια του συμφώνου αυτού, οι οικονομικές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα, οι οικονομικές ρυθμίσεις, έλεγαν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ποσοστό ελλείμματος το οποίο μπορεί το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει το επίπεδο των επενδύσεων και δεν μπορεί να υπάρξει, να γίνει δεκτός προϋπολογισμός ο οποίος δεν σέβεται το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Συνεπώς λοιπόν η Ουγγαρία δεν είναι μόνη ε, όταν δημιουργεί μια αρχή η οποία ελέγχει το δημοσιονομικό κομμάτι και ιδιαίτερα μετά από αυτά τα οποία εμείς βρισκόμαστε στο στάδιο να εφεύρουμε, προσπαθούμε στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης αφαιρούμε την κυριαρχία των Εθνικών Κοινοβουλίων στον προϋπολογισμό τους. Στην ουσία δεν ξέρω αν η Ουγγαρία έκανε κάτι το οποίο θα έλεγα μπορεί να λειτουργεί προληπτικά, το έκανε πριν τους το ζητήσουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και μία έκθεση πρωτοβουλίας ε, για την επίπτωση της κοινοβουλευτικής κυριαρχίας στον προϋπολογισμό σε σχέση ε, με το τι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ χειρότερο από αυτό που κάνουν οι Ούγγροι. Όπως είπατε αυτό είναι... Δεν πρέπει να βιαστούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς την ουσία του θέματος. Αλλά ο στόχος μας είναι να ελέγξουμε κατά πόσο είμαστε σύμφωνοι ή όχι σε σχέση με τα σημεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με το σχέδιό μας για τα έγγραφα εργασίας. Εκ των προτέρων πριν από την επίσκεψή μας και εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά την χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Η κυρία Γκάλ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να προσθέσω. Να προσθέσω δύο σχόλια για τα πρακτικά. Δεν θέλω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά θα εξεταστούν και θα έχουμε και κάποιες ε, έγγραφες ε, απαντήσεις. Δεν είχαμε τον καιρό να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες. Ένα θέμα είναι αυτό για τους λεγόμενους κύριους ή κέριους νόμους. Υπάρχουν πιο πολλοί τέτοιου είδους νόμοι, λιγότεροι τέτοιοι νόμοι από ότι μετά... Λιγότεροι τώρα από ό,τι πριν από την συνταγματική αλλαγή. Αυτό λοιπόν το θέμα των κέριων νόμων, των κομβικών νόμων, δεν θεωρήθηκε πρόβλημα στο παρελθόν, γιατί ξαφνικά γίνεται πρόβλημα όταν ο αριθμός αυτών των νόμων είναι ο ίδιος ή λιγότερος και μάλιστα οι διεθνείς φορείς είπαν ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους ε, κομβικοί νόμοι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου. Είπαν ότι τέτοιοι νόμοι εξασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου, αλλά τελικά ο αριθμός αυτών των νόμων δεν, δεν αυξήθηκε. Επίσης, αναφέρθηκε το θέμα της μη εκπεφρασμένης κατάρρησης της θανατικής ποινής. <clears throat> Υπάρχει όμως μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία εξακολουθεί να ισχύει και αυτό, αυτή η απαγόρευση θανατικής ποινής παραμένει στο Σύνταγμα και υπάρχουν πολλές συμβάσεις που η Ουγγαρία έχει υπογράψει και το Σύνταγμα μας λέει ότι η Ουγγαρία πρέπει να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της ε, στο διεθνές επίπεδο η Ουγγαρία. Βέβαια το να υπάρχει να υπάρχουν ισόβια δεσμά χωρίς δυνατότητα ε, αναθεώρησης αυτής της ποινή μπορεί να είναι θέμα, αλλά υπήρξανε πάνω από 900.000 άτομα τα οποία ζήτησαν να υπάρχει αυτή η παράγραφος η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα μιας ποινή ισοβίων δεσμών τα οποία δεν επιδέχονται αναθεώρηση. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα βέβαια που χρειάζονται διευκρίνηση γιατί υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να δώσουμε τις, ε, τα σχόλιά μας για τα θέματα αυτά. Κυρία Γκönς. Πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις γιατί θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ε, μου έκανε εντύπωση που υπήρξε παράπονο για τον αριθμό αυτών των νόμων. Δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι το, με, το, με το σύστημα το καινούργιο πλέον έχουμε έναν ε, νόμο συνταγματικό. Επομένως, στο μέλλον δεν θα υπάρχει η ελευθερία και το δικαίωμα της κάθε κυβέρνησης, κάθε μελλοντική κυβέρνησης να πάρει αποφάσεις για την οικογενειακή πολιτική, για τη φορολογία και το καθεξής. Και αυτοί οι κέρι ε, νόμοι ε, ισχύουν και πλέον χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία. Μετά είναι και ο, ο ρόλος ε, των ε, δημόσιων διαβουλεύσεων. Είχαμε κάποια στοιχεία εδώ πέρα, αλλά αν συγκρίνετε τα ερωτήματα ε, τα οποία κλείθηκαν να απαντήσουν οι άνθρωποι με το πραγματικό περιεχόμενο των νόμων υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν, ήταν, δεν κατέστη πολλέ σαφέ τι έγινε με αυτά τα ερωτηματολόγια. Και αν δείτε τι θα σας πούνε για την ποιότητα των δημόσιων διαβουλεύσεων, όχι τα στατικαστικά στοιχεία, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Την επόμενη εβδομάδα μας θα έχουμε περισσότερο χρόνο. κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι είδου συζήτηση θέλουμε να κάνουμε εδώ σήμερα. Ε, δεν θα κάνουμε σήμερα το έργο ε, που μας περιμένει την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε επί του εγγράφου εργασίας που έχει υποβληθεί. Θα ήταν καλό οι Ούγγροι συνάδελφοι ε, να μείνουν σε αυτό το πεδίο λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ όλους για την ποιότητα των εγγράφων. Ναι, γιατί άκουσα κάποιες παρεμβάσεις και ε, μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα για το αντικείμενο της σημερινής συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι τα κείμενα είναι ε, πολύ σωστά, θέτουν κάποια ερωτήματα χωρίς όμως να κάνουν το έργο που θέλουν να κάνουν την άλλη εβδομάδα. Δύο παρατηρήσεις. Έχω και ένα ερώτημα. Αν γνωρίζω καλά τον συνάδελφο Ταβάρες, αξιοποίησε το γεγονό ότι υπήρξε κοινοποίηση ε, κάποιων ε, νόμων οι οποίοι μεταφράστηκαν κιόλας θα ήταν καλό το σύνολο των αντιπροσωπιών να έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα έγγραφα. Γιατί αλλιώς ε, δεν υπάρχει ίση μεταχείριση. Και δεν ξεκινάμε επίση όρει το εγχείρημα τη επόμενη εβδομάδα. Και αυτό συνδέεται με τη συνέχεια. Ε, απλώς ε, με δυσκόλεψε η έλλειψη αυτών των ε, κειμένων και δεν μπορούμε να εργαστούμε χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας ε, αυτά τα ουγγρικά κείμενα. Ζητώ συγγνώμη από τους Ούγγρους συναδέλφους, ε, δεν μιλώ την ουγγρική γλώσσα, με τα βίας μιλώ αγγλικά. Είμαι 100% Γαλλίδα λοιπόν ως προς αυτό. Εγώ θα εργαστώ επί δύο ζητημάτων που με προβληματίζουν. το ζήτημα της ε, ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, γιατί υπήρξαν ε, μεταρρυθμίσεις σε αυτό το τομέα που δημιούργησαν κάποια ερωτηματικά. Και δεύτερον, για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις μεγάλες ε, τροποποιήσεις στον εργασιακό κώδικα. Αν κατάλαβα καλά, θα έχουμε το, την επόμενη εβδομάδα το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεών μα, γιατί πρέπει πραγματικά να έρθουμε σε επαφή με τι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά όλοι είμαστε υπέρμαχοι της ε, προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν είναι μόνο ε, αστικά ή πολιτικά δικαιώματα αλλά και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Θα σταματήσω εδώ γιατί πρέπει να μείνουμε στο ε, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστούμε κυρία Σίπελ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εργαστεί για αυτά τα κείμενα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τα έχουμε αυτά πρωτού πάμε στην Ουγγαρία επιτόπου. Και θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια βάση πραγματικών στοιχείων σε σχέση με τα θέματα αυτά ως βάση συζήτησης. Το ερώτημα βέβαια τίθεται αν συμφωνούμε με αυτά τα έγγραφα ή όχι, αλλά είναι φανερό πόσο δύσκολο είναι να αντικατοπτρίσει κανείς όχι μονάχα με μονομένα στοιχεία, είναι δύσκολο να εξετάσει κανείς εξονυχιστικά όλα τα άρθρα του χάρη για τον νόμο περί μέσων ενημέρωσης και δεν αρκεί να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία μεμονωμένα, πρέπει να δούμε και το σύνολο, ποιο είναι το συνολικό αποτέλεσμα και αυτό ίσως ισχύει και για άλλα νομοθετήματα. Νομίζω ότι το θέμα της ε, του κατά πόσο συνάδουν με το δίκαιο όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, έχουμε αποφάσεις κοινοβουλίων και τα, του Κοινοβουλίου του Ουγγρικού. Τα κοινοβούλια είναι ακρογωνία η λύθη της δημοκρατίας μας και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά αυτά τα οποία αποφασίζει ένα κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά, το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε ένα ερώτημα μπορεί πολλές φορές να έχει και μία επιρροή στην απάντηση που μας δίνεται. Επομένω, είναι ένα δύσκολο θέμα. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι επειδή είναι μικρή η παρουσία των μελών εδώ αυτό δείχνει μικρό ενδιαφέρον, μάλλον αντανακλά το γεγονό ότι είναι πέμπτη απόγευμα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε εν καιρό να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση για θέμα αυτό και ελπίζω ότι οι προσπάθειε οι οποίε έχουν γίνει θα μα βοηθήσουν και σε άλλε περιπτώσει παρά το γεγονό ότι ελπίζω ότι δεν θα προκύψουν τέτοιε περιπτώσει στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Προβληματίζομαι λίγο ε, τι ακριβώς θα κάνουμε, θα ελέγξουμε τα 27 συντάγματα των 27 κρατών μελών με την εντολή που έχουμε λάβει. Θα είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό ε, πνευματικό εγχείρημα. Με τα χαράς ε, θα ήθελα να το αναλάβω, αλλά νομίζω ότι εδώ μιλάμε μόνο για την Ουγγαρία και δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι νόμιμη αυτή η, αυτό το εγχείρημα. Ε, βασικός πυρήνας του εγχειρήματο είναι το κράτος δικαίου. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό διαδικαστικό στοιχείο. Μπορεί να συμφωνώ, να διαφωνώ με κάποια από τους ουσιαστικά ζητήματα κράτους δικαίου σε αυτό το έγγραφο εργασίας, αλλά για... σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, οι νόμοι πρέπει να είναι προβλέψιμοι, σίγουροι. Και ο πρόεδρος αυτό που είπε στην αρχή της συνεδρίας, ότι ε, αυτή η αντιπροσωπεία, η αποστολή στην ε, Ουγγαρία, βρίσκεται εκτός δικαίου σε ό,τι αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να διευκρινίσουμε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαφωτίσει ε, την Ουγγαρία για ζητήματα κράτους δικαίου, με τα χαράς και να δεχτούμε όλες αυτές τις διακρινήσεις. Αλλά να μας πείτε τι ακριβώς κάνουμε και ποια είναι η νομική βάση για αυτό το εγχείρημα και για το, τη σημερινή συνεδρίαση και για το έγγραφο εργασία και για την επόμενη την αποστολή ad hoc στην Ουγγαρία την επόμενη εβδομάδα. Γιατί επιλέγουμε αυτά τα ζητήματα που βεβαίως ε, με τα χαράς να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων των ε, όλων αυτών των εργαζομένων που εργάζονται υπό άθλιες ε, συνθήκες στα εργοστάσια εκεί. Αλλά γιατί αυτούς τους τομείς συγκεκριμένα. Κάτι άλλο η χρονική συγκυρία δεν είναι και καλύτερη. Στι 20 Σεπτεμβρίου έχουμε. Είναι μαύρη ημέρα στην ιστορία της Ουγγαρίας. Έξι χρόνια πριν, στις 20 Σεπτεμβρίου, υπήρξε, ε, υπήρξαν μαζικές βιοπραγίες της αστυνομίας στους δρόμους της Βουδαπέστης. Εκατοντάδες άνθρωποι ε, κακοποιήθηκαν βάναυσα από την αστυνομία Εκατοντάδες άνθρωποι που αποδείχθηκε ότι ήταν αθώοι φυλακίστηκαν από την ε, ε, κυβέρνηση που εκπροσωπείται εδώ σήμερα ε, στο Προεδρείο της Επιτροπής από την κυρία Γκόγκς και θα ήταν καταπληκτική ιδέα αυτή την ημέρα να ακούσουμε και μια συγγνώμη επιτέλους. Διακόπτη ο Πρόεδρος έχετε, θίγεται αυτό το ζήτημα κάθε φορά που παίρνετε το λόγο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Είπατε ότι εδώ μιλάμε για το κράτος δικαίου. Το θέμα είναι ότι έχει λάβει εντολή η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ από το Κοινοβούλιο να αποσταλεί αντιπροσωπεία εφόσον έχει αποφασιστεί με απόφαση πλειοψηφίας να αποσταλεί μια αντιπροσωπεία οπουδήποτε, στη Γερμανία, στην Ισπανία, την Ελλανδία, όπου και να είναι αυτό, αυτή η αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει. Το θέμα είναι ότι έχει αποσταλεί αυτή την προσωπία στην Ουγγαρία γιατί αυτό αποφάσισε με εντελώς δημοκρατικό τρόπο το Κοινοβούλιο και γίνεται και είναι μια αντιπροσωπεία ad hoc ε, που ε, περιλαμβάνεται στον διαδικαστικό κανονισμό. Έτσι. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να τα έχετε υπόψη σα ακριβώς για να βοηθήσει αυτή την αντιπροσωπεία να επιτύχει τον στόχο της χωρίς να προκαταλάβει το αποτέλεσμα και τα απορίσματα των συζητήσεων που θα γίνουν στη Βουδαπέστη, αλλά για να βοηθήσει αυτές τις συζητήσεις να έχουν νόημα. Δεν είμαστε εδώ λοιπόν για να κάνουμε μια επισκόπηση όλης της πολιτικής κατάστασης στην Ουγγαρία. Απλώς να δούμε κατά πόσον τα έγγραφα εργασίες είναι έγγραφα τα οποία θα είναι χρήσιμα για τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην εκπόνηση της τελικής έκθεσης που θα συντάξει ο εισηγητής μας. Και η κυρία νομίζω ότι πρέπει να λάβει το λόγο σαν τελευταία πρωτού επανέλθουμε στον κύριο Ταβάρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσά και το Ρουί Ταβάρη για το έργο σας στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου που μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο. Νομίζω δεν θα πρέπει να βάλουμε το άρωτρο πριν από το άλογο, όπως λέμε στην Ιρλανδία. Θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μετά από την επίσκεψή μας στην Ιρλανδία και όχι πριν. Ακόμα και στο έγγραφο που παρουσιάστηκε τα γεγονότα είναι ανοιχτά σε διαμφισβήτηση και διαφορετικές ερμηνείες. Εγώ κατανοώ λοιπόν όλους αυτούς όλοι αυτοί με του οποίου θα μιλήσουμε στην Ουγγαρία θα έχουν ίσω διαφορετικέ οπτικέ γωνίε και ερμηνείε και θα διαμφισβητήσουν κάποια στοιχεία σε αυτό το έγγραφο εργασία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο αυτό το έγγραφο, μα δίνει ένα πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο για τα πράγματα στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μα. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ένα ανοιχτό πνεύμα στο διάλογο αυτό με την Ουγγρική κυβέρνηση και να διατηρήσουμε καλή θέληση από όλες τις πλευρές αν θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ξέρω ότι πρέπει να μην πάρουμε βεβαιασμένε αποφάσει, να μην καταλήξουμε σε κρίση πρωτού δούμε τα στοιχεία, δεν θα πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την έκθεση και τι διαδικασίε αυτέ και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην παραβιάσουμε την κυριαρχικότητα κρατών μελών. Κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το σεβόμαστε. Πρέπει λοιπόν να πάμε στην Ουγγαρία και να πάμε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, εγώ έρχομαι από μια χώρα η οποία έχει υπερηφάνεια, νιώθει υπερηφάνεια γιατί δεν έχει γραπτό Σύνταγμα. Τα συντάγματα λοιπόν ποικίλουν από χώρα σε χώρα και πρέπει να κρατήσουμε ένα ανοιχτό πνεύμα συζητήσεις μας. Ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι θέμα ουσίας. Όλα αυτά καθορίζονται όμως από ορισμένα δεσμευτικά θα έλεγα στοιχεία από τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία περιλαμβάνει και την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Όλα τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και το δικό σας και το δικό μου, όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από κάποιους δεσμευτικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνουν τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η πρώτη, το πρώτο άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ζητά την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στην επίσκεψή μας στη Βουγαπέστη. Κάποιοι από εμάς θα είναι μέλη αυτής της αντιπροσωπείας και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταβάρης πλέον για να κλείσει το θέμα αυτό τελευταίο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ και τους Κιώδης, ιδιαίτερα τους Ούγκρους συναδέλφους που έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει. και γιατί έχετε τα γλωσσικά μέσα να γνωρίζετε τα πράγματα. Όχι μόνο από αυτό βέβαια, πάντως η συνδρομή σας είναι καλοδεχούμενη και πολύτιμη. Σημείωσα αυτά που είπατε και θα προσπαθήσω να τα εντάξω στην προσπάθεια που κάνω. Υπάρχουν ορισμένα σημεία λοιπόν, τα οποία σύντομα θα σχολιάσω. Ευχαριστώ τον Άλμπερτ. Τον Φρανκ, για την προσπάθεια, για την συνεισφορά του. Να πω ότι έτσι και αλλιώ το σύμφωνο αυτό ε, δεν είναι η συνθήκη ευρωπαϊκή και δεν ξέρω ακριβώς βέβαια ποια είναι τα δικαιώματα τα αποκλειστικά του Κοινοβουλίου στον δημοσιονομικό τομέα στη δική μου χώρα αλλά γι' αυτό ακριβώς έτσι και αλλιώ το σύμφωνο αυτό ε, δεν περιλαμβάνεται ε, στην εκθεσή μου γιατί δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί αλλά δεν πάει να παραμένει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Για τους, Για τους νόμους εγώ χαιρετίζω τα σχόλια της Κίνγκα Γκάλ και των άλλων συναδέλφων Νομίζω ότι το θέμα... Το θέμα δεν είναι ο αριθμός των ε, κομβικών ε, νόμων, αλλά η ταυτόχρονη έγκριση πολλών τέτοιων νόμων μαζί με το Σύνταγμα και αν αυτό έχει ένα αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός παράλληλου συντάγματος. Δεν καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα στο θέμα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα θέματα τα οποία μπορεί να τεθεί. Επίσης θα θέλαμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση με τον πληθυσμό. Κατανοώ και αυτά τα οποία λέχθηκαν και από τις ε, δύο πλευράς. Άμα τα στείλετε γράφος μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο κείμενό μας. Η αίτηση της ε, κυρίας Βερζιά νομίζω ότι έχουν ε, κάθε νόημα. Οι μεταφρασμένες τα μεταφρασμένα κείμενα που έχουμε είναι τα ίδια με αυτά που έχει η Κομισιόν και ίσως η Γραμματεία μπορεί να μας τα δώσει. Αυτά που έχει η Επιτροπή μας, μάλλον η Γραμματεία τα έχει. Είναι χρήσιμο όλοι να έχουν τα ίδια κείμενα εργασίας και για τα έγγραφα εργασίας. Νομίζω ότι πρέπει να συναντηθούμε μετά από την επίσκεψη στη Βουδαπέστη για να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για το περιεχόμενο των εγγράφων εργασίας και αυτά που λέτε λοιπόν για την παιδεία και το, τους εργασιακούς νόμους. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές λοιπόν και αυτά τα έγγραφα εργασίας, αν συμφωνήσουν όλοι, μπορούν να είναι και βάση για αίτηση γνωμοδότησης από άλλες επιτροπές όπως την Επιτροπή Απασχόληση, η Επιτροπή συνταγματικών θεμάτων. Για να κλείσω, δεν πρόκειται να ελέγξουμε 27 συντάγματα, ακόμα και άγραφα συντάγματα που άντε να τα ελέγξει κανείς. Απλώς ε, εξετάζουμε τις ε, πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία της Ουγγαρίας ε, όλα τα κοινοβούλια έχουν συνταγματική κυριαρχία και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο επίσης. Δεν πρέπει να τύχει παραβίαση σε αυτή η κυριαρχικότητα των κοινοβουλίων, ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι' αυτό μας εξελέξανε. Όλοι οι ευρωβουλευτές ως ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν την δημοκρατική κυριαρχία του δικού μας οργάνου να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπερεθνική κυριαρχία είναι επέκταση εθνικής κυριαρχίας. Όλα αυτά δεν είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε εδώ πέρα σε μεταφυσικό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Να προσθέσω ακόμα ότι την επόμενη εβδομάδα η αντιπροσωπεία μας εξακολουθεί να είναι μια ερευνητικού χαρακτήρα αποστολής. Μια ερευνητική των πραγματών αποστολή και αυτός είναι ο στόχος της. Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά όταν λέμε ότι είναι απλώ μια ερευνητική των πραγματών αποστολή και αυτό περιμένουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρε. ευχαριστώ όλα τα μέλη τα οποία συνέβαλαν στην εμπλουτιστική συζήτηση για το έγγραφο εργασία και αυτού που προσπαθούν να βοηθήσουν στη σύνταξη των εγγράφων εργασία. Κάποιοι από εμά θα είμαστε ιδιαίτερα εμπεπλεγμένοι στην επίσκεψή μα στη Βουδαπέστη και φυσικά θα κάνουμε μια αναφορά στο σύνολο τη Επιτροπή μα μέσω του εισηγητού μα. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε όλου και για σήμερα αυτά είχαμε. Θα τα ξαναπούμε.